Good morning, colleagues, um, and we can... Uh, Καλημέρα, συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι ήδη εδώ. Τμήμα του πακέτου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα κοιτάξουμε το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων. Η Τάνα Φαγιών είναι η συγκέντρια και θα τη δώσουμε το λόγο για 5 λεπτά. Στη συνέχεια θα πάρουμε το λόγο και οι σκιώδει. Η Τάνια έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κλόντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω λίγο παραπάνω από 5 λεπτά. Ελπίζω όμω όχι πολύ παραπάνω. Και θα εξηγήσω αυτά που θα ρωτήσουν ενδεχομένω οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ που μου δίνετε λοιπόν το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ύπαρξη των, ε, του χώρου εσωτερικών συνόρων χωρίς έλεγχο είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Το Σέγγεν είναι από τα πια επτά επιτεύγματα τόσο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσο και για τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα δημορφωθεί το μέλλον του Σέγγεν. Η σωστή λειτουργία του χώρου Σέγγεν θα πρέπει να συνοδεύεται και από έναν αριθμό πολιτικών σε ό,τι αφορά την διάσκηση των συνόρων, σε ό,τι αφορά και επίσης από χρηματοδοτικά μέσα για την εφαρμογή όλων των πολιτικών αυτών. Αφενός λοιπόν το Σέγγεν βοηθά τους πολίτες μας να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να συμμετέχουν και στην ε, ενιαία αγορά και επιπλέον επιτρέπει την προστασία των εξωτερικών συνόρων καθώς και του χώρου Σέγγεν. Ως εισηγήτρια καλωσορίζω επίσης και το μέσο χρηματοδότησης που θα μετα φέρει όλες αυτές τις πολιτικές στην πράξη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των θεωρήσεων, των συνόρων. Σε 7 χρόνια θα έχουμε περίπου 10 δις ευρώ και μιλάμε για πενταπλάσια ουσιαστικά αύξηση σε σχέση με το τρέχον ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων τα τελευταία 7 χρόνια που έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο κοινό ευρωπαϊκό έργο. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε απάντηση σε αυτές τις νέες προκλήσεις και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια σειρά μέτρων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα. Θα θυμάστε άλλωστε και την εισαγωγή των συστηματικών ελέγχων και των βάσεων δεδομένων σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά σύνορα και την εκτοφυλακή. Επίσης υπάρχει και ένα καινούργιο σύστημα, το EES και το EPS, αλλά η εμπιστοσύνη παρόλα αυτά δεν έχει ανακτηθεί 100%. Πολλά κράτη-μέλη επιμένουν να συνεχίζουν τους εσωτερικούς ελέγχους συνόρων παρά το γεγονός ότι εμείς επιμένουμε ότι δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Αντί για συνεργασία βλέπουμε με έναν απομονωτισμό. Και αυτό... Και αυτό γιατί στις χώρες αυτές πάντα οι λαϊκιστές είναι αυτοί που καταλήγουν στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα λυπηρό γεγονός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επικεντρωθώ σε κάποια θέματα λοιπόν σήμερα. Βασικός σκοπός της διαχείρισης των συνόρων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για ενοποιημένη διαχείριση θεωρήσεων και συνόρων. Αυτά τα μέτρα πάντα θα πρέπει να ορίζονται με σαφή τρόπο και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να πετύχουμε σωστή προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και προστασία της ελευθερής κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω ότι επικεντρώνονται υπερβολικά στις ε, πτυχές της ασφάλειας και λιγότερο στις πτυχές της καλύτερης διαχείρισης μεταναστευτικών ροών. Δεν υπάρχει λοιπόν επικέντρωση στη διευκόλυνση διάσχεσης των σύνορων για ταξιδιώτες ε, οι οποίοι ταξιδεύουν καλή πίστη και δεν αποτελούν κανένα κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική για τις θεωρήσεις επίσης θα χρηματοδοτηθεί από το εργαλείο αυτό και αποτελεί πραγματικά κλειδί για την οικονομία, τον πολιτισμό. Και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πολιτική για τις θεωρήσεις και γι' αυτό πρότεινα ένα ελάχιστο κατόφλι για τη χρηματοδότηση. Οποιοδήποτε στόχο θέτουμε θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη χρηματοδότηση. Ιδάλω δεν μπορεί να μεταφραστεί σε δράσει. Σε ό,τι αφορά τι συγκεκριμένε πολιτικέ και τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών, θα πρέπει να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αποφύγουμε και γι' αυτό λοιπόν το αναπτύσσω το θέμα αυτό στην έκθεσή μου. Έχουμε νέες τεχνολογίες τώρα και γι' αυτό πρότεινα μία ειδική προσθήκη σε ό,τι αφορά τη διάταξη που θα αποτρέπει την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμελητών δικαιωμάτων για την προσωπική σφαίρα και τα προσωπικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τα τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει προστασία από διακριτική μεταχείριση. Τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν άλλωστε τα μέσα αυτά για να χρηματοδοτήσουν ε, μέτρα στα εξωτερικά σύνορα, αλλά και για να ελέγξουν τα θαλάσσια σύνορά τους. Θα πρέπει να αναφέρουμε αποστολές διάσωσης στη θάλασσα, όπου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, και τις ε, αρχές αυτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν δικλείδες ασφαλείας και σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιώματων αυτών και του διεθνούς δικαίου. Το εργαλείο αυτό θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε επίσης μέτρα στα, στους hot spots ε, και σε ό,τι αφορά τις Διαδικασίε των σύνορων. Θα πρέπει να σεβαστούμε σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα της ε, διεθνή προσδιαγραφή για τους διεθνούς, ε, για τους ζητούντες άσυλο και για τα άτομα που χρήζουν βοήθεια. Να διευκολύνουμε επίσης ε, το πέρασμα των σύνορων για τους ταξιδιώτες καλή και αν εγκρίνουμε το μέτρο αυτό θα σώσουμε παράλληλα και πολλές ζωές στην Μεσόγειο. Στο πλαίσιο λοιπόν του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και η ανάπτυξη ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματος για ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός να απομακρυνθούμε από τα κέντρα που ξεφορτώνουμε κόσμο και θα πρέπει να εστιαστούμε σε θετικέ πράξεις, να μεταφραστούν όλα αυτά σε θετικέ πράξεις. Οι ανθρωπιστικές λοιπόν θεωρήσεις θα ήταν ένα τέτοιο μέτρο. Τέλος, να πω δύο λόγια για τα μέσα που αφορούν τρίτα κράτη. Έχουμε μία σειρά μηχανισμών που μπορούν να εφαρμοστούν υπό τέτοιου όρου. Τα μέτρα αυτά λοιπόν θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένα και να έχουμε και κάποιες ασφ... δικλείδες ασφαλείας για να χρηματοδοτήσουμε μέσα κατεπίγουσας ανάγκης. Τέλος, να επισημάνω ότι χρειάζεται σωστή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών προκειμένου να υπάρξει δημοκρατική επισκόπηση. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει στις διαδικασίες προετοιμασίας των προγραμμάτων αυτών, των θεματικών εργαλείων με πράξεις κατά εξουσιοδότηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει τη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω και στην μελλοντική συνεργασία με όλους τους κοιόδης και με την Επιτροπή και αν έχετε ερωτήσει. ευχαριστώ να σας απαντήσω. E Ευχαριστώ. Ο Κάρλο Κουέλιο έχει το λόγο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Τάνια Φαγιόν για το έργο της. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Το ΕΛΚ θα υποβάλει τροπολογίες που θα αντικατοπτρίζουν τη θέση του, αλλά ως αφετηρία θα ήθελα να πω ποιε είναι οι βασικέ μα ανησυχίε σε σχέση με το σχέδιο έκθεση. Πρώτον, δεν πιστεύουμε ότι ο κανονισμό αυτό θα πρέπει να προβλέπει οποιαδήποτε χρηματοδότηση για κάτι που δεν υπάρχει ούτε, ε, ούτε προγραμματίζεται να υπάρξει. Νομίζω ότι συμφωνεί η συγγήτρια μαζί μου, γιατί έχετε διαγράψει όλες τις αναφορές σε νέα ε, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα πληροφόρησης η χρηματοδότηση θα πρέπει να κατευθυνθεί μόνο στην, ε, σε υπάρχοντα συστήματα και σε εκείνα που θα έχουν εγκριθεί έως ότου τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Για τους ίδιους λόγους, για ποιο λόγο να προβλέπετε χρηματοδότηση για ενωσιακές ανθρωποστικές ε, θεωρήσεις. Δεν μπορούμε να, να τις επιβάλλουμε αυτές στα κράτη-μέλη. Εμείς ως Κοινοβούλιο μπορούμε στην καλύτερη περίπτωση να εκδώσουμε κάποια σύσταση για ένα τέτοιο μηχανισμό και παρόλα αυτά εσείς θέλετε να προβλέπετε χρηματοδότηση. Εμείς διαφωνούμε. Δεύτερον, βεβαίως είμαστε υπέρ μιας ε, ολοκληρωμένης προσέγγισης. Να εξετάζει κανείς ένα πρόβλημα με όλα του τα στοιχεία και να προσπαθεί να βρει συνολικές λύσεις. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναμαγνύουμε τους μηχανισμούς χρηματοδότησης. όσα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του Ταμείου Ασύλου θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από εκεί. Και όσα σχετίζονται με τα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα. Το να αναμειγνύει αυτά δεν είναι καλή πολιτική, ούτε είναι και κάτι εφικτό με βάση το δημοσιονομικό κανονισμό. Παρ' όλα αυτά, σε ευχαριστώ Τάνια για την έκθεσή σου και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για το ECR, ο κύριος Βίστανσεν. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για το έργο της. Ωστόσο, ε, η δική μας πολιτική γραμμή είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που έχει υιοθετήσει η εισηγήτρια. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι αφαλές και ανεύθυνο ε, να ισχυρίζεται κανείς ότι η μεγάλη πλειοψηφία που διέρχεται από τα εξωτερικά σύνορά μας είναι ε, bona fide ταξιδιώτες που δεν ε, συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια της Ένωσης συνολικά. Αυτό δεν ισχύει. Ε, παρά, το γεγον, παρά τα όσα λέγονται εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι και μη ρεαλιστική και επικίνδυνη. Στην παράγραφο 3, για παράδειγμα, η εισηγήτρια αποσυνδέει τον έλεγχο των συνόρων με την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων εντό της Ένωσης, ε, αφαιρώντα την, την λέξη, τον όρο προπόθεση. Μήπω θα έπρεπε να μα εξηγήσει η εισηγήτρια το σκεπτικό τη, γιατί με βάση τα όσα είπα και νωρίτερα, η εσωτερική ασφάλεια και η ελευθερία κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς, βεβαίω ε, εξαρτάται από το αν έχει κανείς ε, ασφαλή εξωτερικά σύνορα. Υπάρχει και η τροπολογία 23, όπου η συγγήτρια ε, αφαιρεί την δυνατότητα να χρησιμοποιείται τελωνικός εξοπλισμός και για τους ε, συνοριακούς ελέγχους, για λόγους ασφαλείας. Μα αυτό θα βοηθούσε την συνεργασία, όπως ακριβώς αναφέρεται και στην πρόταση Κομισιόν. Ποιο είναι το πρόβλημα ε, με το να καταθήσουμε το Ταμείο πιο αποτελεσματικό. Επίσης, διαφωνούμε με το γεγονός, με την άποψη της ε, εισηγήτριας ότι θα πρέπει να χρηματοδοτείται η έκδοση ανθρωπιστικών θεωρήσεων και οποιοδήποτε αντίστοιχο μηχανισμού ανθρωπιστικών θεωρήσεων στο μέλλον, που θα θεσπιστεί στο μέλλον, όπως είπε και το ΕΛΚ. Χωρί να θέλω να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε, είναι σαφέ ότι η δική μα προσέγγιση είναι αντίθετη με εκείνη τη εισηγήτρια θα πρέπει προτεραιότητα να είναι η διαχείριση των συνόρων, ιδίω η πρόληψη και ο εντοπισμό τη παράνομη μετανάστευση και του διασυνορικού εγκλήματο. Επίση, στόχο του κανονισμού είναι η συνεργασία στον τομέα τη έκδοση ε, χορηγήσεων για να διευκολύνονται τα ταξίδια ε, χωρίς ελέγχους. Αυτοί οι δύο στόχοι λοιπόν ε, της Κομισιόν μέσω του κανονισμού θα έπρεπε να είναι και οι στόχοι ε, της έκθεσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Ένωση. Επίσης θεωρώ ότι είναι κρίσιμο ο μηχανισμός να μπορεί να υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με τρίτες χώρες. Από αυτή την άποψη ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να... Ε, ε, ασχολείται μόνο με την, τον εντοπισμό, την πρόληψη ε, και την σύλληψη εκείνων που ε, προβαίνουν σε παράνομες διελεύσεις των συνόρων, αλλά θα πρέπει να προβλέπει και τη χρηματοδότηση των σταθμών αποβίβασης, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ. Μπόντιλ Βαλέρο για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, βάλτε τα ακουστικά σας. Ε, πρέπει να πω ότι εγώ σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με την κυρία Φαγιόν. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε ε, υπερβολικά στην ασφάλεια. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι αφελές ή ανεύθυνο το ε, να προβλέπεται ανθρωπιστική ε, θεώρηση. Πρέπει να αποτελεί ε, τμήμα αυτής της δουλειάς. Έχουμε εργαστεί επί αυτού του θέματος εδώ στο Κοινοβούλιο επί μακρόν. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση και η διαδικασία αυτή. Βεβαίως η ψηφοφορία επίκειται στο άμεσο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει με ικανοποιητικό τρόπο και τις δικές μας σκέψεις και απόψεις ε, θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε την έκθεση αυτή με τροπολογίες, αλλά στην κατεύθυνση ενίσχυσης ε, της έκθεσης που έχει συντάξει η Τάνια. Δεν νομίζω ότι θα είναι εφικτό να ανερθούν όλοι οι έλεγχοι που γίνονται στα εσωτερικά σύνορα, γιατί υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τα κράτη-μέλη. Λέω απλώ ότι η ίδια η έκθεση δεν πρόκειται να επιτύχει το στόχο αυτό. Ακριβώ γιατί υπάρχουν και άλλε διαστάσει που πρέπει να συνεκτιμήσει κανεί. Και είμαι πεπισμένη ότι τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να διενεργούν ε, εσωτερικού ελέγχου για αρκετό διάστημα. Εγώ, ξέρετε, κατάγομαι από μια χώρα ε, και, ε, όπου γίνονται τέτοιοι έλεγχοι και ξέρω ότι γίνονται τέτοιοι έλεγχοι και στην γέφυρα ορεσούν. Και διαφωνώ. Αλλά είναι προφανέ ότι μέσω μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν όλοι οι εσωτερικοί σύνολοι. Να πω κάτι για αυτό που είπε ο κύριο Βίστησεν. Όταν, είπατε, ε, για την, ε, όταν μιλήσατε για ε, παράνομη μετανάσταση, νο, νόμιζα ότι είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα τον χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Δεν υπάρχει παράνομη μετανάστευση. Κάτι παράνομο είναι κάτι που αντιτίθεται στην νομοθεσία. Ναι, μπορεί η μετανάστευση σε ορισμένε περιπτώσει να αντιβαίνει στου κανόνε. Άρα είναι μια παράτυπη μετανάστευση, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον, ε, τον όρο παράνομη μετανάστευση. Και απογοητεύομαι γιατί νόμιζα ότι είχαμε σημειώσει κάποια πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα. Πρόεδρο. Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν την έχουμε σημειώσει την πρόοδο αυτή. Τάνια, θέλεις να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν. Ωραία, παρακαλώ πολύ σύντομα και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία ε, και να ευχαριστήσω και την κυρία Φαγιόν για την έκθεσή της. Είναι μια έκθεση που βασίζεται σε μεγάλο έργο. Κάποια σημεία που πρέπει να, στα οποία πρέπει να αναφερθώ. Ένα πολιτικό. Πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και της ε, διευκόλυνσης των ε, ροών στα σύνορα. Στα σύνορα διέλευσης. Είναι σημαντικό να προστατευτεί η ασφάλεια και εμείς θεωρούμε ότι η έκθεση επιτυχάνει έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό ισορροπίας. Κάποια τεχνικά ζητήματα. Η έκθεση ε, προτείνει ότι θα πρέπει ε, να ε, επιτυχάνονται αυτά μέσω κατευθυνσιοδότηση πράξης. Ε, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να είναι ευέλικτος και ταχείας αντίδρασης. Η έκθεση αναφέρεται στην αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από το 75% στο 85%. Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα μέσα αυτά είναι τα μέσα που προτείνουν ε, τη μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν αρκετέ δυνατότητες ε, συγχρηματοδότηση, ακόμα και για 85, 90 και 100%. Ε, το 75% είναι 25% πάνω από τα διαρθρωτικά ταμεία. Όσον αφορά τι πληρωμέ και τι ενδιάμεσε αξιολογήσει, 30%. Νομίζω ότι αυτό προτείνει η συγκήτρια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υψηλό. Ε, μπορεί αυτό να μην είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσά, αλλά πρέπει να το συνυπολογίσετε και αυτό. Γιατί η ενδιάμεση αξιολόγηση θα γίνει το 2024 ε, με βάση στα όσα ε, θα έχουν γίνει το 21, 22 και 23. Θυμηθείτε ότι όσον αφορά τις πληρωμές ή την εκτέλεση αν θέλετε, τα ταμεία αυτά θα εκπνεύσουν το 2029. Το 2023 λοιπόν δεν είναι στην πραγματικότητα το μέσο της ε, διάρκειας της περίοδου εφαρμογής. Βρίσκεται στην αρχή ακόμα. Γι' αυτό ε, από άποψη χρηματοδότησης βρισκόμαστε στο μέσο, το, 2023 είναι, στο, είναι το μέσο της περίοδου, αλλά από άποψη εκτέλεσης όχι για, την, για το 30% για ελάχιστο ποσοστό για την κοινή στρατηγική ε, πολιτική θεωρήσεων, εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό της συγκέντριας. Θέλω όμως να πω ότι ο τομέας των θεωρήσεων είναι εκείνος όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ε, όσον αφορά την εφαρμογή τους στην, στα τρέχοντα ταμεία. Και τα λέω αυτά γιατί αυτά ισχύουν και τα τρία ταμεία, γιατί παρόμοιες ε, τροπολογίες έχουν κατατεθεί και για τα τρία μέσα. Όσον αφορά την ανάμειξη των δραστηριοτήτων, εγώ έχω εξηγήσει και στο παρελθόν ότι αυτό είναι μια δυνατότητα, όχι υποχρέωση. Και τέλος, να πω όσον αφορά την παράνομη και παράτυπη μετανάστευση, εμείς στην πρότασή μας χρησιμοποιούμε τον όρο παράνομη, ε, γιατί αυτό αντικατοπτρίζει, αυτό αντικατοπτρίζει και την, την συνθήκη. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία. Τέλος, συνεργασία με τρίτες χώρες. Υπάρχει ένας περιορισμός 2%. Είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στο τρέχον μέσο, αλλά είναι πολύ σημαντικό αν θέλετε το γεγονός ότι έχουμε κατά νου ότι η συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι πάρα πολύ ε, σημαντική και για τους σκοπούς που θέλει να εξυπηρετήσει η κυρία ε, Φαγιόν για τη διέλευση, την απρόσκοπτη διέλευση των συνόρων για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται να υπάρχει καλή διαχείριση των, των ροών ταξιδιωτών, μεταναστών στα σύνορα. Γενικά, πάντως, διαφωνούμε με την λογική των ε, ποσοστών συνολικά. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Um... Σας ευχαριστώ πολύ για να είναι πραγματικά ξεκάθαρα τα πράγματα, να φέρετε σύντομα στην ε, συνθήκη και η θέση του Κοινοβουλίου είναι πως πρόκειται για παράτυπη και όχι παράνομη μετανάσταση. Δεν είσαι παράνομος παρά μόνο όταν ε, κριθείς ως παράνομος. Ε, μπαίνεις, ε, ε, ελέγχεσαι και μετά ορίζεσαι ως παράνομος ή παράτυπο. Εδώ στο Κοινοβούλιο είσαι παράτυπο. Αυτό ισχύει εδώ και 10 χρόνια, οπότε πρέπει να είναι σαφές. Όχι, δεν υπάρχει θέμα και τίποτα, δεν υπάρχει διαδικαστικό. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, συγγνώμη, δηλώνω ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου ότι πρόκειται για παράτυπους μετανάστες. Η κυρία Βαλέρο τεχνικός έχει δίκιο. Ναι, τεχνικός κύριε Πρόεδρε, δεν το αφισβητώ αυτό. Απλώς σας ζητώ να μου στείλετε την νομική βάση αυτού. Κάποια στιγμή ακούστε μας πριν να μας κρίνετε και να πείτε πως δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Παρακαλώ πείτε μου πού τα λέει όλα αυτά, πού τα λέει, ε, πού, ποια είναι η νομική βάση. Κοιτάξτε κύριε Βίστησεν, είπα μόλις πως η Κομισιόν δηλώνει αυτό που είναι στην ε, συνθήκη. Είπα στη συνθήκη πως εν συντομία αναφέρεται στη συνθήκη και η θέση του Κοινοβουλίου ε, είναι εδώ και 10 χρόνια ότι θέλουμε να μιλάμε για παράτυπη μετανάστευση. Κανείς δεν είναι παράνομος μέχρι ότου έτσι κρυθεί από την ίδια την, από την ε, εδώ, εφόσον έχει έρθει πια εδώ. Καταλάβατε ποια είναι η θέση. Συγγνώμη που λίγο θύμωσα. Ξέχασα ε, ότι η κυρία Βαγιών πρέπει και να απαντήσει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς για να το συζητήσουμε. Ε, άλλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας διευκρινίσατε μια ακόμη φορά ποια είναι η σωστή ορολογία και για τους υπόλοιπους να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές, τους κοιόδης ε, την Κομισιόν για τις παρατηρήσεις. Ε, φυσικά και θα τις λάβω υπόψη. Στόχος μου είναι να βρούμε σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και τη διευκόλυνση νόμιμης διέλευσης και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε την καλύτερη δυνατή συμβιβαστική ε, λύση. Σας ευχαριστώ όλους πολύ και η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 1η Δεκεμβρίου. Προχωράμε στο επόμενο σημείο. Τι κάνατε, εσείς αντικαθιστάτε την κυρία Χολμάγερ, μάλιστα. Επόμενο σημείο είναι η εξέταση του σχεδίου έκθεσης της Μόνικας Χολμάγερ. Ο κύριος Μπέκερ θα πάρει τη θέση της, σας ευχαριστούμε. Και έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστούμε κυρία Μπέκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλήσω γερμανικά για να παρουσιάσω την ε, τοποθέτηση της κυρίας Χόλμαϊρ, η οποία δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ. Καταρχάς, η, η συγγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσταση. Η πρόταση αποτελεί μια εξαιρετική βάση για τις μελλοντικές μας εργασίες. Τώρα, να κοιτάξουμε στα σημεία επικέντρωσης της εισηγητρίας σε ό,τι αφορά το σχέδιο της ε, έκθεσης για τη θέσπιση ενός Ταμείου Ιστορικής Ασφάλειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει διάφορες υποχρεώσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα αποτελέσματα ερευνών του όλα για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα σταλίες, μέχρι και απάτε σε ό,τι αφορά το ESF, θα πρέπει να διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, οι ετήσιες εκθέσεις απόδοσης ε, θα πρέπει να διαβιβάζονται αυτόματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο υπό σύνοψή, ε, αλλά και σε, στην πλήρη του έκταση, αν ζητηθεί, προκειμένου οι νομοθέτε να μπορούν να αξιολογούν την εφαρμογή του προγράμματος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν πιο πολύ ευελιξία, γιατί υπάρχει διαφορετικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων αυτών. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, αναφέρεται ελάχιστες δαπάνες αναστόχο. Και το σχέδιο έκθεσης προβλέπει, για παράδειγμα, αύξηση του ανώτατου ορίου για τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων και πιο ευέλικτη διαμόρφωση των ανώτερων ε, ορίων για τη δημιουργία, για παράδειγμα, υπόδομων, μεταφορών και το καθεξής. Αν τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίζουν από μόνα τους τα σημεία προτεραιότητάς τους, η επένδυση στην καταπολέμηση της, του κυβερνού εγκλήματος και την αντιμετώπιση τέτοιων άλλων εγκλήματων θα πρέπει να λάβει κίνητρα. Να υπάρξουν κίνητρα λοιπόν για μέτρα στον τομέα αυτό. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πιο παντώνη αιρεσιμότητα. Στο άρθρο 13 κοιτάμε την χορηγήση της δεύτερης δόσης ε, σε ύψος 30% των ε, συνολικών ταμείων. Θα πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση όμως ό,τι αφορά τη δεύτερη δόση αυτή τα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει επίσης να προσαρμόζονται. Η σημασία συνεργασίας με τα τρίτα κράτη λαμβάνεται υπόψη και έτσι στην έκθεση δεν υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά την σύγκριση με τα κράτη-μέλη. Για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δράση για τα κράτη-μέλη και να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα, προβλέπεται να μπουν τα εκτελεστικά αυτά μέτρα στο διδακτικό του κειμένου, προκειμένου να μπορεί να είναι σωστά οργανωμένη η εφαρμογή, θα πρέπει να ψηφιστούν ξεχωριστά τα θέματα αυτά σε σχέση με τις θεματικές διευκολύνσεις. Για να υπάρχει λοιπόν τώρα καλύτερη αξιολόγηση Ορίζονται κάποιοι τομεί, όπω, ε, για παράδειγμα δείκτε. προστίθενται κάποιοι δείκτε. και δύο λόγια για την μετέπειτα διαδικασία δεδομένων των παρόμοιων δομών με άλλες δομές, η Ευρωπαϊκή η Συγγήτρια προτείνει να υπάρξει συνεργασία με τις εισηγήτριες για το άσυλο και το Ταμείο Μετανάστευσης και με το Ταμείο Διαχείρισης Θεωρήσεων και Συνόρων. Υπάρχει κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την αξιολόγηση και τις υποχρεώσεις αναφοράς. Επίσης, να υπάρχουν εναρμονισμένα χρονοδιαγράμματα στο, στην Επιτροπή. Η εισηγήτρια προσβλέπει στη συνεργασία με τους σκιώδεις και ανυπομονεί να ακούσει τα σχόλιά σας. Να σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much, Mr. and thank you again for... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέικερ και ευχαριστώ που αντικαθιστάτε την κυρία Χολμάιερ. Θα προχωράμε με αυτόν τον το σημαντικό φάκελο λοιπόν. Και τώρα η Σεσίλ, εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο που μας έδωσε την πρόταση ε, αλλαγής της συναδέλφου Χολμάγερ. Εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε σε ένα κλίμα μέγιστης συνεργασίας για αυτό το θέμα της ασφάλειας που διαρκώς εξελίσσεται και απαιτεί ε, ισχυρή και συντονισμένη απάντηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πλευράς όλων των κρατών μελών δηλαδή. Επαναλαμβάνω μια βασική αρχή ε, βασική για την δική μου πολιτική ομάδα, είναι ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, μπορούμε να το πετύχουμε μόνο, όχι μόνο με τα μέτρα αντιπαράθεσης, αλλά και με τα μέτρα πρόληψης. Πέρα, ε, κάποιες από τις τροπολογίες που εγώ θα υποβάλω εξ ονόματος της ομάδας μου ε, των σοσιαλιστών. Ε, οι τροπολογίες λοιπόν που θα υποβάλω θα θα επιμείνουν ε, στην πρόληψη και θα προπονητήρουμε και συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα για να αξιολογήσουμε τα βαθύτερα αίτια, κυρίως ε, για το θέμα που αφορά την ριζοσπαστικοποίηση και άρα την ενίσχυση των πολιτικών ε, πρόληψης, κυρίως από πλευράς ευαίσθητων, ευάλωτων ανθρώπων. Η εισηγήτρια αφήνει ένα περιθώριο δράση σχετικά ευρύ στα κρατημέλη όσον αφορά τι δράσει που θα πρέπει να αναλάβουν. Εμεί ομάδα θεωρούμε ότι η ευελιξία απαραίτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με την διαφάνεια και την ε, ε, κατανομή των πόρων ε, και άρα θα πρέπει να είναι και σύμμορφη με στόχους που με το στόχο της σαφήνειας και της διαφάνειας. Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε δράσης. Αυτό σημαίνει στο πλαίσιο ενός Ταμείου Οικονομικής Στήριξης θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, καταβολή πόρων σε όσους δεν ε, σέβονται τους ε, ελάχιστους κανόνες για αυτό το τομέα. Η πρόταση για την ε, παραβίαση του κράτους δικαίου ε, εξετάζεται σε αυτή την Επιτροπή και είμαι βεβαία ότι θα βρούμε ενδιαφέρουσε απαντήσεις στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν την εισηγήτρια και είμαι βεβαία ότι θα φτιάξουμε μια σωστή σχέση συνεργασίας για το εγγύς μέλλον και σας ευχαριστώ. Thank you very much, And for who else have? Um... Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Σεσίλα. Επόμενος, Η υπόλοιποι σκιώδεις. Κύριος Φρανς, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Καταρχήν, τα πράγματα βαίνουν σε σωστή κατεύθυνση. Η ερώτηση μου αφορά το άρθρο 3. Εκεί διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ή μάλλον διαπιστώνω ότι γίνεται λόγος για μέτρα και όχι για ε, προθέσεις γιατί και έργα για ποιο λόγο έγινε αυτή η αλλαγή επίσης γίνεται αναφορά στην ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Νομίζω ότι θα πρέπει όμω να εξειδικεύεται και κατά θέμα αυτή η κατεύθυνση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση αντιρατσιστικών προγραμμάτων στην αστυνομία, εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχει μια τέτοια γενικόλογη αναφορά. Θα ήθελα να εξειδικεύεται σε μορφές ρατσισμού, αλλά και την επεξεργασία της ε, εθνικοσοσιαλιστικής ιστορίας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να προβλέπετε ε, εξειδικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και λόγω των εξελίξεων που έχουν στην Ευρώπη. Επίσης, σημαντικό είναι και η καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Και πολύ θετική ε, θεωρώ την αναφορά για τα μέτρα για τους πληροφοριοδότες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά στον αφορά του σκιώδεις. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Ωραία, η Κομισιόν τότε. Όχι, ε. Κύριε Μπέκερ, θέλετε να πείτε κάτι ε, στο τέλος της συζήτησης. Όχι. Λοιπόν, προθεσμία για την ε, κατάθεση τροπολογιών είναι η 6η Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκερ για άλλη μια φορά για το γεγονός ότι ε, εκπροσωπήσατε εδώ την κυρία Χολμάιερ. Πάμε στο σημείο 12, το οποίο όμως χρειάστηκε να αναβληθεί για λόγους ενωτέρας βίας. Οπότε θα διακόψουμε τώρα. Διακόπτουμε για 10 λεπτά και ξαναρχίζουμε στις 10. Because, um, because point 12 has had to be postponed. For... Επειδή αναβάλαμε το 12. The rapporteur has asked for the postponement. So we postpone until 10 o'clock. Ο εισηγητής συζήτησε να αναβληθεί. Σταματάμε λοιπόν μέχρι τις 10. Ζητώ συγγνώμη.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 Uh, Συνάδελφοι, να σας ενημερώσω για κάτι. Ε, περιμένουμε την κυρία Ντάλη, που είναι στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ε, έχουν ψηφοφορία. Τελειώνει όμως. Γι' αυτό σας παρακαλώ να περιμένουμε λίγα ακόμη λεπτά, να τελειώσει και να έρθει. Συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, ε, σημαντικές ψηφοφορίες σε άλλες επιτροπές, είναι συντονίστρια. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν, ε, αλλά με έχουν ενημερώσει ότι θα έρθει σύντομα. Okay, colleagues, uh, for your patience. Um, Ευχαριστώ συνάδελφοι που περιμένατε υπομονητικά. Ευχαριστούμε Μίριαμ που έτρεξες να έρθεις εδώ. Ξέρετε, έχουμε συντονιστές και συναδέλφους που είναι πολύ δραστήριοι και σε άλλες επιτροπές σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Λοιπόν, πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Ζητώ και εγώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την κατανόησή σας. Θα προσπαθήσω να συνέλθω από το τρέξιμο, αλλά η παρουσίασή μου θα είναι η ίδια. Είναι λίγο σαν το strictly come dancing, ε. Τρέχει ο ένας από εδώ, τρέχει ο άλλος από εκεί. Να πω ότι μιλάμε για το σχέδιο έκθεσης, για την πρόταση για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, που είναι ένα από τα ε, τομεακά προγράμματα που εμπίπτουν και εντάσσονται στο επόμενο πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Ντάλη, ως εισηγήτρια για το ταμείο αυτό, υπό το επόμενο ΠΔΠ, θα ήθελα να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις της. Να ξεκινήσω λοιπόν με την αρχή της αλληλεγγύης και του ίσου επιμερισμού των ευθυνών, την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, τη δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης, την προώθηση ε, της ε, κοινωνικής ένταξης και την ε, ενισχυμένη βιωσιμότητα ε, της ε, πολιτικής μετανάστευσης. Προφανώς το θέμα της μετανάστευσης δεν μπορεί να εναπόκειται μόνο σε κάποια, σε κάποια εξωτερικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα γιατί δεν αφορά μόνο τα κράτη-μέλη. Είναι κοινή πρόκληση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έλεγα επίσης ότι είναι και παγκόσμια η πρόκληση αυτή. Σκοπός του Ταμείου Ασύλου μετανάστευση είναι να υπάρχει ένας προπολογισμό 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ε, ασχολείται με τις προκλήσεις που απορρέουν από τη μετανάστευση. Ως ε, ε, εισηγήτρια θεωρώ ότι το Ταμείο αυτό ανταποκρίνεται στις ε, ανάγκες προκειμένου να υποστηριχθούν τα μέτρα και οι δράσεις των κρατών μιλών για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μετανάστευσης και τις νομικές τους υποχρεώσεις. Εγώ, ξέρετε, κατάγομαι από την ε, Μάλτα. Είμαστε χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων που περνούν τη Μεσόγειο και καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι ε, μια ε, χώρα μόνη τη να διαχειρίζεται τέτοιε μεταναστευτικές ροέ. και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επιδεικνύεται αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όταν αντιμετωπίζουν τέτοιε καταστάσεις. Κεντρικό σημείο της έκθεσής μου είναι η εισαγωγή ελάχιστων ποσοστών για κάθε στόχο και υπό τα εθνικά προγράμματα και υπό την ε, θεματική διευκόλυνση. Και κάθε, ένας από του στόχους που αναφέρεται στο άρθρο 3 θα πρέπει να δέχεται 20% χρηματοδότηση. Ξέρουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θέλουν μια κάποια ευελιξία όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων, ωστόσο πιστεύω ότι η ευελιξία αυτή δεν θα πρέπει να πλήττει την επίτευξη των διαφόρων στόχων. Η ευελιξία θα πρέπει να συνδέεται με μέτρα που θα εξασφαλίζουν την, τον δίκαιο επιμερισμό των πόρων και τη διαφάνεια όσον αφορά τις ενωσιακές δαπάνες. Επιπλέον, ε, θέλω να υπάρξει ανώτητα, ανώτατο όριο 5% για τη χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων. Πιστεύω ότι ε, η ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να κατευθύνεται κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη και στις δράσεις τους. Και αυτό ε, αντικατοπτρίζεται και στις τροπολογίες μου. Χρειαζόμαστε συστήματα υποδοχής, επαρκή και συστήματα εξασφάλισης ε, δυνατοτήτων για την δίκαιη μεταχείριση, ιδίως για τους ε, ασυνόδους ανηλίκους και τους πρόσφυγες ε, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Και παρά το γεγονός ότι το Ταμείο αυτό καλύπτεται από τον κανονισμό κοινών διατάξεων, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι πιο εξειδικευμένοι κανόνες. Θα πρέπει να υπάρχει εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, κάτι που θα πρέπει να υποστηριχθεί. Επίσης, προτείνεται νέο άρθρο για την ε, ε, εμπλοκή αυτών των αρχών. Επίσης, ε, υπάρχουν και διεθνείς οργανώσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει τα κράτη-μέλη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων πρέπει να, να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών που άλλωστε είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Επίσης, έχω υποβάλει τροπολογία για τον τίτλο του κανονισμού, ώστε για άλλη μια φορά να περιλαμβάνει και την κοινωνική ένταξη και όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς αρκετοί δρόμοι ασφαλού μετανάστευσης, ιδίως για εκείνου που χρειάζονται προστασία. Και ε, καλό τα κράτη-μέλη να διερευνήσουν όλες τις, εξετα... τις ε, πιθανές επιλογές ε, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια. Επίση, ένα λειτουργικό σύστημα χρειάζεται και μια ε, βιώσιμη πολιτική επιστροφών που θα πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε εκείνους που χρήζουν διεθνούς προστασίας και ταυτόχρονα να επιστρέφουμε εκείνους που δεν έχουν δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο ε, υποχρεώσεις είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργικότητα ενός οποιοδήποτε συστήματος ασύλου αυτή η επιστροφή μπορεί να χρηματοδοτείται από το Ταμείο. Όπως εξήγησα νωρίτερα, θα πρέπει ε, ε, να, να υπάρχει για αυτό το τομέα ανώτατο όριο 5%. Επίσης, χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου αυτού, πρέπει να χρηματοδοτούνται ε, και εξωτερικές δράσεις, αλλά θα πρέπει να συνάδουν πάντοτε με την εξωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος θέλω να επισημάνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του για την λογοδοσία της Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των κονδυλίων στη βάση συγκεκριμένων συγκριτικών δικτών και της αξιολο... της αλλά και τις αιτήσει εκθέσεις που θα ε, συντάσσονται. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους χιώδεις, στις παρατηρήσεις τους και με επικοδομητικό πνεύμα θα προχωρήσουμε στην, ε, στο έργο αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Περνάμε στους ε, σκιώδεις. Ο κύριος Κοέλιο από το ΕΛΚ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή ο κύριος Λένας ε, βρίσκεται σε μια σημαντική ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, για το κλίμα, για το περιβάλλον αυτή τη στιγμή, έχω την τιμή να μιλήσω εξ ονόματός του σχετικά με την έκθεση της κυρίας Ντάλη. Ο κύριος Λένερ ευχαριστεί την κυρία Ντάλη για την εργασία της μέχρι τώρα και ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο ε, εργάστηκε με ε, όλους. Ε, το κείμενο είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας. Ο κ. Λένερ συμφωνεί με την εισηγήτρια να συμπεριληφθεί η αλληλεγγύη και η δίκαιη μοιρασιά των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη-μέλη ως στόχο του Ταμείου. Ε, αυτή τη στιγμή κάποια κράτη-μέλη φαίνεται να απομακρύνονται από αυτή την αρχή, ενώ η αλληλεγγύη είναι το, η ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και ε, μετανάστευση. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να τονιστεί και να τονιστεί ως συγκεκριμένο στόχος του Ταμείου. Επιπλέον, ο κύριος Λένας καλωσορίζει την θέση της συγγήτριας για ε, μια κλίδα κατανομής για τα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιστροφή των παράτυπων μεταναστών μάλλον παράνομων μεταναστών, είπε ο μιλητή, όπου αυτό χρειάζεται. Να, στηριχθεί, λοιπόν, ε, να στηριχθούν οι επιστροφέ, όπως ε, ήδη στηρίζει και η Επιτροπή. Εν γέννη, η Κομισιόν έχει υποβάλει μια δίκαιη και ισορροπημένη πρόταση για την κατανομή των πόρων και αυτή η ισορροπία θα πρέπει να διατηρηθεί σε σχέση με την αντιμετώπιση μελλοντικών ε, προκλήσεων είναι σημαντικό αυτό το πλαίσιο να ε, περιέχει αρκετή ευελιξία. Γι' αυτό ο κ. Λένατ δεν θεωρεί πως η προτινόμενη εισαγωγή ελάχιστων επιπέδων ε, δαπανών για τους διάφορους στόχους του Ταμείου είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Θεωρεί πως το σύστημα θα πρέπει να προβλέπει στόχους με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία κάθε φορά καλωσορίζει τη ιδέα της τροπολογίας της συγκήτριας για την αυστηρή, ε, αυστηρό κανονισμό για τη χρηματοδότηση τρίτων χωρών. Εφόσον τώρα όμως ε, ε, διερευνώνται οι δυνατότητες για αυξημένη συνεργασία στην περιοχή, δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση σε γειτονικέ τρίτες χώρες μόνο. Αντίθετα, θα πρέπει χώρες και άλλες χώρες να είναι επιλέξιμες όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση της κρίσης της μετανάστευσης. Για όλα αυτά τα θέματα, ο κ. Λένα το προσβλέπει σε καρποφόρα ε, συνεργασία με την κυρία Ντάλη, τους υπόλοιπους ε, σκιώδες και όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η σιαρ η είναι η Κριστίνα Λούνμπεργκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές. Όσον αφορά αυτό το ταμείο, βλέπουμε σημαντική αύξηση και πώς θα πρέπει να καταναμηθεί αυτό το ταμείο. Θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια. Αυτό το νούμερο 40% για τις επαναπατρισμούς θα πρέπει να αυξηθεί και άλλο γιατί θεωρούμε πως πολλοί κόσμος έχει φτάσει με παράνομο τρόπο ε, στις χώρες μας, ιδιαίτερα στην ε, Σουηδία, τη χώρα μου, χρειαζόμαστε δέσμευση μεγαλύτερη ε, για τη βοήθεια προς τους, βοήθεια μάλλον σε σχέση με τους επαναπατρισμούς. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τρόποι για να φτάσει κανείς νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι ποσοστός, υπάρχουν οι οδηγίες, θα, πρέπει, θα έπρεπε κανείς να μπορεί να φτάσει πιο ε, εύκολα. Εδώ πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το Ταμείο για την ένταξη των ανθρώπων που φτάνουν εδώ, ώστε να μπορούν όντως να ενταχθούν στην κοινωνία με καλύτερο τρόπο. Ε, ε, αυτά λοιπόν και αυτή είναι η δική μου άποψη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω πως έχουμε άλλον σκιώδη παρόντα εδώ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Η Σεσίλ Κέγγε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Μυριάμ για την παρουσίαση αυτού του ταμείου που είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ήθελα να παρέμβω για ορισμένα σημεία που θεωρώ πως έχουν προτεραιότητα. Βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι αρκετά περίπλοκη και ευαίσθητη. Πολλά κράτη-μέλη αντί να αυξάνουν τις πολιτικές μετανάστευσης ή να εφαρμόζουν ή να διαθέτουν ε, ταμεία για τις πολιτικές ε, ένταξεις ε, περικόπτουν και μειώνουν. Εγώ πιστεύω πως αυτό το ταμείο και μέσω αυτού του ταμείου θα μπορέσουμε να καταστήσουμε κατανοητό πως η μείωση από πλευρά των κρατών μελών αυτού του ταμείου θα έπρεπε να σημαίνει και άμεση πρόσβαση για τις τοπικές ε, αρχές που ασχολούνται με τη μετανάστευση. Γιατί αν εξαρτώνται μόνο από τα κονδύλια που φτάνουν στα κρατημέλη, αυτό θέτει ε, σε κίνδυνο την πολιτική ένταξη ε, επιτόπου. Πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε γιατί είναι αυτή η κατάσταση σε πολλές χώρες όπου καλές πρακτικές που ήδη είχαν θεσπιστεί σταματούν ή κάνουν και πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να δημιουργούμε ανθρώπους που ζουν αόρατοι, ζουν παράτυπα και έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε όσον αφορά την ασφάλεια. Δημιουργείται μια κατάσταση ανασφάλειας. Η άλλη μου παρατήρηση αφορά τις πολιτικές επαναπατρισμού. Εγώ επιμένω και λέω ότι η επιστροφή ένας άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει αλλά με αξιοπρέπεια. Ποτέ δεν πρέπει να συγχαίουμε τις πολιτικές επιστροφής με τις, τα αίτια των ε, για το από έχουν ε, φύγει αυτοί οι άνθρωποι. Προγράμματα ένταξη τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης θα πρέπει να γίνονται. Ε, πιστεύω πως αν προσπαθήσουμε να το τονίσουμε όλα αυτά θα ενισχύσουμε περισσότερο αυτό το σημείο. τέλο. αν μου επιτρέπει, Μίριαμ, το γεγονός είναι ότι πολλές από αυτέ τι πολιτικέ ένταξει. Ε, συχνά ε, ε, φτιάχνονται από το Υπουργείο Εξωτερικού με την οπτική της ασφάλειας. Γιατί να μην ζητήσουμε από τα κατημέλη να φτιάξουν το καθένα Υπουργείο που να ασχολείται με τη διαχείριση των κονδυλίων και των στρατηγικών για την ένταξη αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλ. Μίριαμ, θέλεις τώρα εσύ να μας πεις τα απορίσματά σου. 6 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η κυρία Ντάλη, ευχαριστώ τους σκιώδεις και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους για την έκθεσή μου. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, η πρώτη αφορά το, ε, κανονισμό του Δουβλίνου και το άρθρο 17 που ορίζει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης ε, όπως φαίνεται στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά εδώ θα ήθελα να κάνουμε τροπολογίες ότι αναδικατοπίζεται η θέση του Κοινοβουλίου. Και εδώ θέλω να καλέσω τους κοιόδης για να υπογράψουν αυτά Αυτέ οι τροπολογίε. Η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά τα παραρτήματα. Πολλέ τροπολογίες έχουν κατατεθεί για να εξασφαλίσουμε ότι είναι σύμμορφε με το πνεύμα των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί για τον κανονισμό αυτό και θεωρώ πως τα παραρτήματα είναι η καρδιά αυτού του κανονισμού. και προσβλέπω σε καλύτερη συνεργασία, περισσότερη μάλλον συνεργασία με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 6 Δεκεμβρίου. Η Κομισιόν ζητά το λόγο. Έχουμε ψηφοφορίε όμω. Παρακαλώ να είστε πάρα, πάρα πολύ σύντομοι. Κοιτάξτε, σα ε, κουνάω το χέρι μου εδώ και ώρα, αλλά δεν με είδατε. Θα είμαι πολύ σύντομο να αναγνωρίσουμε τη τεράστιο έργο της ηγήτριας, να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Η αλληλεγγύη είναι μέσα στην πρόταση του, της Κομισιόν. Αυτός είναι ένας από τους στόχους. Καταλαβαίνουμε ε, την πρόταση για την αλληλεγγύη ως έναν επιπλέον στόχο, αλλά θα πρέπει να είναι Ε, ο μόνος στόχος ε, οι κατηγορίες επανεγκατάστασης ή μετεγκατάστασης αλλάζουν. <coughs> Δεν μπορούμε λοιπόν μονίμως να το βάλουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Εξωτερική διάσταση. Καταλαβαίνω τους στόχους της εισηγήτριας, ωστόσο θα πρέπει να θυμόμαστε πως κάνουμε πολλά για τη σωστή εφαρμογή αυτών των πολιτικών και χρειάζεται ένα εξωτερικό συστατικό ε, για την επανένταξη των επιστροφών, να βοηθήσουμε τις ίδιες χώρες να φτάσουν σε ένα επίπεδο προστασίας επίσης. Χρειαζόμαστε παραπάνω από 5%. Ε, και τέλος, για να κλείσω με αυτό, Πρόεδρε, όπως είπα και νωρίτερα, και για την κυρία Ντάλη, το κατόφλι που έχουμε επιβάλει εδώ και η αύξηση του επίπεδου συγχρηματοδότησης μπορεί να είναι κάπως υπερβολικό γιατί είναι το μέσο με το υψηλότερο ε, ποσοστό συγχρηματοδότησης. Έχουμε εδώ περιλάβει τη δυνατότητα 100%, 90% και 75% και τελευταία παρατήρηση αφορά τα μίνιμουμ ποσοστά 20-20-20. Όπως είπε ο κύριος Κοέλιο, οι ανάγκες αλλάζουν. Δεν είναι οι ίδιες ούτε για όλα τα κράτη, ούτε για όλους τους στόχους. Οπότε το 20% για όλους είναι ένα, δεν, δεν είναι πολύ καλό ε, μέτρο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Μίριαμ. Συνάδελφοι, λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Και Έχουμε εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Εισηγητή έχει έρθει, θα πάρει τώρα το λόγο. Κύριε Κοράου, θέλετε το λόγο, όχι. Ωραία, περνάμε λοιπόν τότε στην ψηφοφορία. Ελεκτρονικά. Colleagues, eh, who, can you just indicate if you don't have your electronic card? Συνάδελφοι, ναι, έχετε φέρει τις κάρτες σας. Έχω την αίσθηση ότι Αυτές οι μέρες είναι δύσκολες. Τι κάνετε με την κάρτα σας όμως. Κανες άλλος έχει πρόβλημα με την κάρτα του. Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 12. Έναρξε. Είναι ακόμα ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 46 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Πέρασε. Εγκρίνεται. 50. 50, 51, 8, 53, 54, 56. Ταυτόσημε. Έναρξη. Πέρα. Εγκρίνεται. Εννέα υπέρ. Ε, έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Μάλλον ναι, έναξη ψηφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Η 10. Ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. 61. εξε. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Έναρξη. πέρασε. Εγκρίνεται. 71. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. 72. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 73. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 74. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 76. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Έτρωγικές σκέψεις. 13. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκαπέντε. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία ένα. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Έναρξη. Πέρας. Πέρας. 19. Έναρξη. Πέρας. Πέρας. 20. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Έναρξη. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Οι δύο ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Τι δύο. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Έναρξε. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Πέρας. Εγκρίνεται. 26-27 ταυτόσημες. Ψηφίζουμε. Πέρας κρίνεται. 28. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 29. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 30. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 32. Έναρξε. Πέρας. Απορρίπτεται. 4 και 35 ταυτόσημες. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 5. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 40. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Το κείμενο αποστροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται 30 ψήφοι. 34 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στον συγητή. Και τώρα περνάμε σε μία ε, ψηφοφορία για τα δικαιώματα των μεσοφιλικών ατόμων. Ε, ερώτηση ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευρεία συνένεση. Εγκρίθηκαν στις 19 Νοεμβρίου και με email αποστάλει η ερώτηση στις 20 Νοεμβρίου. Συζητήθηκε από την διάσκεψη των Προέδρων και θα περάσει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 128. Περνάμε λοιπόν στην ε, μία και μόνη ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 30 ψήφοι υπέρ, 7 κατά καμία αποχή. Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Ευχαριστώ για την ε, υπομονή σας σήμερα το πρωί και για τις καθυστερήσεις που είχαμε ζητώ συγγνώμη. Συνάδελφοι, ε, θα προχωρήσουμε στο σημείο 16 σε λίγο, μόλις ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Απαλλαγή 2017. Όποιος θέλει να αποχωρήσει, ας το κάνει ησύχως, παρακαλώ. Um, Ωραία. Συνάδελφοι, προχωράμε με τα σημεία της μύρισης διάταξης. Αν θέλετε να φύγετε, κάντε το άλλο σας, παρακαλώ ήσυχα. Σημείο 16 έως 21, 26 με συγχωρείτε, για την απαλλαγή του προπολογισμού Ξεκινάμε με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού των οργανισμών. Θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας για τις 11 αυτές γνωμοδοτήσεις, για, τις, ε, για τους ε, διάφορους οργανισμούς, τον προπολογισμό της Κομισιόν, τους οργανισμούς ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών και του Ευρωπαίου επόπτη προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κύριε Φράνς, παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις γνωματοτήσεις σας. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ως συνήθως αναφέρομαι στα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου και γενικά ε, συμφωνώ με τα συμπεράσματα αυτά το ελεγκτικό συνέδριο επικρίνει το γεγονός ότι ε, πολύ συχνά οι οργανισμοί δεν κοινοποιούν επαρκώς τις ε, θέσεις που προκυρήσουν. Στον Ευρωπαϊκό Επόπτη ε, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, επίσης, ελέγχθηκε μόλις μία πληρωμή το 2017. Υπάρχει πρόβλημα με τις ε, πληρωμές και τον έλεγχό τους. Θα περιοριστώ σε κάποια σημεία κριτική για κάποιους οργανισμούς. Ο οργανισμός ΕΑΖΟ για το άσυλο είναι ο μοναδικός αποκεντρωμένο οργανισμό για τον οποίο ε, δεν συνιστά το ελεγκτικό συνέδριο απαλλαγή. Δεν υπάρχει ακόμα σαφή εικόνα. Ο προϋπολογισμός του 2016 ε, ήδη δεν είχε λάβει, δεν είχε τύχει τη απαλλαγή από το Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι αυτό συνέβη τον Οκτώβριο του 2018 μόλις, διότι υπάρχουν προβλήματα και στις προμήθειες και στο προσωπικό του οργανισμού αυτού. 10,3 του όγκου των πληρωμών ε, χαρακτηρίζονται από το ελληνικό συνέδριο ως μη συμμορφούμενους με τους κανόνες. Παρ' όλα αυτά επισημαίνεται ότι ο οργανισμός έχει λάβει μέτρα και βρίσκεται πλέον σε σωστή κατεύθυνση. Συνάδελφοι, δεν ξέρω αν εσείς θα συμφωνούσατε με την επιλογή για την ΕΑΣΟ. Σε αντίθεση με την ΕΑΖΟ, η Frontex παρουσιάζει ε, διαφορετική και πολύ θετική εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν ε, μεγάλες υπερεκτιμήσεις των αναγκών στον προϋπολογισμό κάτι που οδήγησε σε μη απορρόφηση κονδυλίων και μη, εκτέλεση του, μη αξιοποίηση του ε, προϋπολογισμού. Υπάρχουν προβλήματα και για την συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Και κάτι τελευταίο. Παρά το γεγονός ότι το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ο οργανισμός ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν έχει ε, ικανούς πόρους προσωπικού, και οικονομικούς για την εκτέλεση των καθηκόντων του δεν υπάρχει δυνατότητα να ε, παρεμβαίνει η κοινωνία των πολιτών. Ε, και έτσι ε, χάνεται η ευκαιρία να ενισχύεται συνολικά η ευρωπαϊκή πολιτική. Τέλος, επικρίνω την ανισορροπία γυναικών ανδρών στα διοικητικά συμβούλια. Μόλις 11 από τα 70 μέλη των οργανισμών είναι γυναίκες. Στα έργα, επίσης, πάντως, γενικά τηρείται το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει μεγάλο ε, πρόβλημα, το γεγονός είναι το γεγονός ότι το 90% των ε, πληροφορικών συστημάτων έχουν ανατεθεί σε τρεις μεγάλες ε, εταιρείες πληροφορικής. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη εξάρτηση και η αδυναμία ενός από τους παρόχους, ενδεχόμενη αδυναμία που θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Πρέπει ο εξοπλισμός να να, γίνεται, να, να, τον προφημιθεύεται ο οργανισμός με διαφανείς κανόνες και με εξασφάλιση της δυνατότητας συμβατότητας με τα συστήματα τρίτων χωρών. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημεία κριτικής τα οποία θέλω εδώ σήμερα να επισημάνω. Νομίζω επίσης συνάδελφοι ότι από κοινού θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για την απαλλαγή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν έχω τη λίστα των σκιωδών. Α, ευχαριστώ μόλις την έλαβα. Να δώσω το λόγο ε, τώρα στους σκιώδεις για την απαλλαγή των διαφόρων οργανισμών. ΕΛΚ, Ρομπέρτα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Φράντς, για την απαλλαγή για όλους αυτούς τους οργανισμούς, όλα τα σχέδια ε, γνωμοδότησης για την απαλλαγή αποτελούν καλή βάση για τις διαπραγματεύσει, για αυτούς τους φακελούς. Εμείς είμαστε υπέρ των περισσότερων από αυτές τι γνωμοδοτήσεις ε, αποτελούν δίκαιη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των οργανισμών στον τομέα του δικαιοσύνη και των εσωτερικών. Συμφωνούμε για περισσότερη διαφάνεια και δημοσιότητα στι θέσει που ανοίγουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωστόσο, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για τα σημεία τα οποία υπάρχουν στις διάφορες γνωμοδοτήσεις. Ας πούμε, για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο εισηγητής καλεί τα κράτη-μέλη να κατανείμουν τη φύση των ποσών στους ετήσιους λογαριασμού στα εθνικά τους προγράμματα ΑΜΕΦ και ISF, γιατί ε, ακόμα μάλλον και αν η σημερινή πρακτική είναι σύμμορφη με τις απαιτήσει. Είναι σημαντικό σημείο που πρέπει να διαβιβάσουμε στους συναδέλφους μας που διαπραγματεύονται το νέο κανονισμό για το νέο PDP μέχρι το 27. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω αν αυτό είναι θέση. Μπορεί μάλλον να περιλαμβάνεται στη γνωμοδότηση που προκύπτει από αυτήν εδώ την Επιτροπή. Και αυτό ειδικά γιατί το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε αυτό του κανονισμού. Το ίδιο και για την γνωμοδότηση για το Eurojust που ζητά ανοιχτή, περιλαμβάνει ανοιχτή σύσταση για το, για το ελεγκτικό συνέδριο που λέει να αναθεωρήσει ε, τον τρόπο με τον οποίο διηρίζονται, μα αυτό δεν το αποφασίζει ο ίδιος ο οργανισμός. Και αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη και όχι από τον οργανισμό. Επιπλέον είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι πόροι που κατανέμονται στον ε, ε, επόπτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχουν αυξηθεί στη διάρκεια των ετών. Είναι σημαντικό να αυξηθούν κι άλλο, αλλά πρέπει να τονίσουμε τις θετικέ κινήσεις του οργανισμού, όπως παρότερη αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο στην έκθεση για την απαλλαγή, για την Europol. Οι αναφορές για την εσωτερική, στην εσωτερική μονάδα παραπομπής δεν ε, είναι σωστές, θα πρέπει να τονίσουμε και να επενήσουμε ε, την εργασία αυτού της μονάδας και όχι να αφισβητήσουμε την νομική βάση για την Ιουνίσα. Η υπεργολαβία για, τα, για την ε, IT ε, έχει ανατεθεί ε, λόγω έλλειψης πόρων. Δεν θα πρέπει επίσης να αμφισβητήσουμε την εντολή της, του οργανισμού αυτού. Δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να περιλαμβάνεται σε μια γνωμοδότηση περί απαλλαγής. Και η παράγραφοι για επιχειρησιακό επίπεδο, η εντολή το Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα είναι σαφή παραδείγματα. Θα στηρίζαμε αυτές τις θέσεις, αλλά μόνο εάν ε, προταθούν στους ε, κατάλληλους ε, φακέλους, όχι στο πλαίσιο της απαλλαγής. Προσβλέπω και την έκθεση, στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για αυτούς τους οργανισμούς για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο σωστή αξιολόγηση για τους οργανισμούς στον τομέα μας. Αυτά και προσλόγω στη συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ, ε, Ρομπέρτα. Από τους σοσιαλιστές η Κατερίνα Τσινίτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κινίτσι, με συγχωρείτε. Να, συναδέλφω, να συγχαρώ ε, τον συνάδελφο για τη δουλειά που έκανε για την απαλλαγή, για τους οργανισμούς γενικότερα και την εργασία που έκανε στους οργανισμούς που ασχολούνται με τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές ε, υποθέσεις και είναι οι οργανισμοί οι οποίοι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τους πιο περίπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή ασφάλεια, μετανάστευση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να ενταχθούν επίσης και να είναι πολύ καλά συντονισμένοι. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η συνάδελφος που μίλησε πριν έκανε κάποιες τέτοιες ε, παρατηρήσεις. Εγώ θέλω να κάνω παρατηρήσεις για την οργανισμό Eurojust που είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός ε, φορέας όσον αφορά το χώρο ε, ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης που θα ανοίξει ακόμη και περισσότερο στο μέλλον λόγω και του αγώνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις ε, ε, για τα διασυνοριακό έγκλημα. Είναι σημαντικό πολύ οι γνωμοδότησεις οι δικές μας αλλά και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήδη καταγράφουν καλύτερη ε, βελτίωση στη διαχείριση ε, της, ε, του σε αυτή. Τώρα, σε σχέση με την Λίζα, είναι βέβαια ένας οργανισμός που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μελλοντικέ προκλήσεις λόγω των πιο περίπλοκων βάσεων δεδομένων, αλλά πάντοτε είναι απαραίτητες αυτές οι βάσεις και βέβαια συμμερίζομαι τους προβληματισμούς του ελεγκτικού συνεδρίου και του συντάκτη για την υπερβολική ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες γιατί είναι μεγάλη εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Ωστόσο δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τόσο είπε η συνάδελφος Μετσόλα γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα πρόβλημα το οποίο οφείλεται στην έλλειψη του ε, προσωπικού. Να σταθώ επίσης τον οργανισμό ΕΑΖΟ. όπου όντω υπήρξαν κάποια ε, προβλήματα διαχείρισης και λογαριασμών στο πρόσφατο παρελθόν. Όμως, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του, της υπηρεσίας για την υποστήριξη στο άσυλο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πτυχές και εδώ αυτό θα πρέπει να μα προβληματίσει όσον αφορά τι αποφάσει που θα λάβουμε. Αυτό ο οργανισμό, κατά τη γνώμη μου, ακολουθεί το σωστό δρόμο για να, για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να καλύψει τα προβλήματα. Καταρχά, ο διορισμό του νέου αντίντερεμ ε, γενικού ε, ε, διευθυντή που έγινε τον περασμένο Ιούνιο δείχνει ακριβώ ότι ο οργανισμός αυτός έχει δεσμευθεί για τι δυνατότητε να να, για να μπορέσει μάλλον πια να παρεμβαίνει και μέσω ενός κατάλληλου συστήματος εσωτερικών ελέγχων. Πιστεύω λοιπόν πως ο οργανισμός είναι στον καλό δρόμο για να ε, απαντήσει στα προβλήματα που είχαν προκύψει και ότι αυτό θα οδηγήσει στην ε, απαλλαγή. Θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή και τους σχιώδεις για να ολοκληρώσουμε την ε, εργασία μας. Πολύ σημαντική ε, λοιπόν είναι η εργασία για την απαλλαγή όλων αυτών των οργανισμών και ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι κρυωμένη και βήχω. Οι σκιώδεις λοιπόν πήραν το λόγο. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Εγώ παρακολούθησα την συνεδρίαση του DGAG. Ήταν μοναδική αυτή η συνεδρίαση, γιατί έχουμε ένα σωρό οργανισμούς που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό ε, το ε, τις παρατηρήσεις ε, και η κυρία Κινίτσι και η κυρία Μετζόλα ε, έδειξαν την υποστήριξή τους, πράγμα που εκτιμούμε. Σε σχέση λοιπόν με την απαλλαγή για το Eurojust, νομίζω πως είναι σωστό που έχουμε χαμηλό προϋπολογισμό σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα είδος διαδικαστικού ρόλου, δηλαδή τη στιγμή που οι άλλοι έχουν ολοκληρώσει τις έρευνές τους και έχουν έναν ε, προϋπολογισμό που να είναι λογικός. Να πω λοιπόν Κατερίνα ότι αυτή η συζήτηση έγινε λεπτομερώς. Οι μεταρρυθμίσεις της ΕΑΣΟ, παρά την έρευνα που γίνεται από την Όλαφ, συνεχίζονται. Ο κύριος ε, Φράντσε έχει κάνει αυτή την επαφή και σίγουρα θα α, ε, μας ενημερώνει. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν συνεχίζονται και είναι απαραίτητες. Ξέρω πως πολλοί συνάδελφοι παρακολουθούν την κατάσταση. Παρακαλώ λοιπόν να συνεχίσετε να παρακολουθείτε κι εσείς, να είμαστε προσεκτικοί. Δεν υπάρχει άλλη επιτροπή που να ασχολείται με τόσε πολλέ ε, υπηρεσίε και οργανισμού. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Κύριε Φραντ, θέλετε να ολοκληρώσετε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για τις παρεμβάσεις τους ε, και τα σημεία αυτά που μας είπατε και προσβλέπω και στην συζήτηση και στην μελλοντική συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λόγκη Πρόεδρος. μία γράφεις τραπολογιών είναι η 6η Δεκεμβρίου. Να πάμε στο σημείο 27 που είναι η παρουσίαση του Μηχανισμού Προτεκτικής Βοήθειας. Ε, η κυρία Βαλέρο είναι η συγγήτρια. Καταφτάνει. Μόλις ε, κάτσε λοιπόν η Μπότλη, μπορούμε να ξεκινήσουμε στο επόμενο θέμα. Okay, I thought I was very early. Και εγώ που νόμιζα ότι είχα φτάσει νωρίς νωρίς. 11 και 10 έλεγε το πρόγραμμα. Yeah, we've up again. Συγγνώμη. Α, ξεκινήσαμε πιο νωρίς. Ευχαριστώ, Μπότιλ. Είχαμε καθυστερήσει λίγο, αλλά τώρα πάμε πιο γρήγορα. Είσαι έτοιμη? Δεν μοιάζομαστε. Να δω αν έχω όλα μου τα χαρτιά εδώ. Ναι, μην βιάζεστε. Παρουσιάζουμε λοιπόν το μηχανισμό πρωταξιακής βοήθειας. Σας σου ειδικά, αν μου επιτρέπετε, βάλτε ακουστικά. Όπω είπατε, πρόκειται για την δημιουργία ενό μηχανισμού πρωταξιακή βοήθεια. Ε, το τρίτο τέτοιο μηχανισμό και μιλάμε για μία σειρά χωρών Κόσοβο, Τουρκία, πρώην Ιεκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και άλλες χώρες, είναι όλες στον κατάλογο. Είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα λοιπόν αυτά. Το σημείο 3 λοιπόν αναφέρει τα Βαλκάνια και τη σχέση με την Τουρκία. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των προηγούμενων ε, μηχανισμών και του τρέχοντος μηχανισμού σε ό,τι αφορά τις χώρες ε, υποένταξη και θα πρέπει να τηρούνται επίσης και οι πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλους τομείς, η κλιματική πολιτική, μετανάστευση και μια πιο ασφαλής Ευρώπη κοιτώντας την ε, πρόταση, το σημείο κίνησής μου. Ήταν να προσπαθήσω να αποφύγω τις επικαλύψεις, να αποφύγουμε επικαλύψεις με άλλα μέσα χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια, αν βρω και που είναι και τα χαρτιά μου, τα βρήκα. Υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα κονδύλια. Τα χρήματα αυτά θέλουμε να βοηθήσουν και στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων με τη μετανάστευση και με την ασφάλεια. Αλλά ήδη έχουμε ένα ενοποιημένο ταμείο για το άσυλο και τη μετανάστευση, για τη διαχείριση των συνόρων την... και επίσης το ταμείο για την βελτιωμένη, την ενισχυμένη εσωτερική ασφάλεια. Άρα εδώ μιλάμε για την πρωτοιαξιακή διαχείριση, για την κοινωνική συνοχή στις χώρες αυτές εδώ θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε και όχι τόσο πολύ στη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης. Προτείνω λοιπόν να αφαιρέσουμε την πτυχή αυτή από το μηχανισμό και να εστιαστούμε ανταυτού στην ενίσχυση των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της αποτελεσματικότητας, της ε, διαχείρισης, ε, προσέγγιση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενίσχυση των ε, κοινωνικών εξελίξεων, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της κοινωνικής ενοποίησης ενίσχυση ε, της περιφερειακής και της συνοριακής επίσης εργασίας. Από πλευρά μου λοιπόν αυτό θα έπρεπε να ένα τέτοιο μηχανισμό. Έκανα λοιπόν σχετικέ ε, προτάσει ε, και τροπολογίε ε, για την έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι επικεντρωνόμαστε λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε στα θέματα διαχείριση συνόρων και διαχείριση μετανάστευση. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να δοθεί μεγαλύτερο βάρο στι άλλε πτυχέ και να συμπεριληφθούν και άλλε ευάλωτε ομάδε όπω η Ρωμά. Και αυτό γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνία στις χώρες αυτές. Και θα πρέπει, θεωρώ, να το κοιτάξουμε αυτό υπό το πρίσμα της κοινωνικής σφαίρας και όχι τόσο πολύ από την ε, οπτική γωνία της διαχείρισης σύνορων να δημιουργηθεί επίσης ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής συμπερίληψης στις χώρες αυτές. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις ε, χώρες αυτές προκειμένου να αναπτύξουν τις αξίες και τις αρχές που εκτιμούμε στην Ευρώπη. Να επικεντρωθούμε επίση στην ε, ενοποίηση και την ενσωμάτωση. Και τελευταίο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και στους νέου μέσω τη εκπαίδευση. Και θα πρέπει να υπάρξει και σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό θα διευκολύνει το έργο μα και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μπόντιλ. Και Ζητάει μία συνάδελφο στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βαλέρο. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το μη πι 3 να γίνει ένα νέο ανεξάρτητο μέσο εντός του νέου ΠΔΠ και να τεθεί σε λειτουργία από το 2021. Αυτό το μέσο είναι μοναδικό και βοηθά με αυτό, με αυτό τρόπο τις χώρες για τις οποίες μιλάμε για την, στην πορεία τους ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προοδευτική τους ανάπτυξη να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, να ενισχυθεί η απόκτηση δεξιοτήτων, η συνεργασία μέσω διασυνοριακών προγραμμάτων και άλλων προγραμμάτων. Και όλα αυτά τα προγράμματα αποτελούν τη βάση των ε, σχέσεων καλής γειτονίας μας, που με τη σειρά της είναι εξαιρετικής σημασίας, ιδίως ε, όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και το διάλογό μας με την Τουρκία. Όλες αυτές οι πτυχές είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτόν τον λόγο προσβλέπω στις μελλοντικέ μας εργασίες. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο, Μπόντιλ, θέλεις να κάνεις κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Α, συγγνώμη, κύριος Νάγκη. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του κύριου Σόγκαρ θα ήθελα να διαβάσω τις ε, παρατηρήσεις του, διότι δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί σήμερα. Θέση του ΕΛΚ είναι ότι η προενταξιακή διαδικασία αποτελεί σημαντικό ε, παράγοντα για την πραγματοποίηση δημοκρατικών και άλλων μεταρρυθμίσεων λόγω του κινήτρου που δίνει η διαδικασία αυτή ε, μέσω της ε, διαδικασίας ένταξης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ε, αποτελεσματική στην προενταξιακή φάση παρά μετά την ένταξη μιας χώρας στην Ένωση. Πέρα λοιπόν από τις διαρθρωτικές οικονομικές, πολιτικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, η συνολική προενταξιδική διαδικασία είναι μια σκληρή διαδικασία από την οποία ε, διέρχονται οι υποψήφιες χώρες και γι' αυτό χρειάζεται ε, αποτελεσματική ε, ενωσιακή χρηματοδότηση η οποία θα μπορεί να ανταποκρίνεται και να δίνει απαντήσεις στις υπάρχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις. Επίσης, υποστηρίζουμε την επικέντρωση της εισηγήτριας στο ζήτημα του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας δικαστικής εξουσίας και της ε, ε, καταπολέμησης της ε, διαφθοράς. Για να ενισχυθούν ε, επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο κ. Σόγκο θα ήθελε να ενισχυθεί η αιρεσιμότητα του προγράμματος προενταξιακής βοήθειας, δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αναστέλει την προενταξιακή βοήθεια σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σοβαρές και μόνιμες παραβιάσεις των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωτών δικαιωμάτων, όπως ε, αυτά καθορίζονται στις δεσμεύσεις που συνάπτονται μεταξύ των υποψηφίων χωρών και της Ένωσης. Λόγω της ταραγμένης ε, πρόσφατης ιστορίας των Δυτικών Βαλκανίων, θέλουμε επίσης να επισημάνουμε την σημασία που έχουν τα μέτρα που θα κατευθύνονται στην ενίσχυση του διαλόγου, ε, τη συμφιλίωση, τον σεβασμό των εθνικών μειονοτήτων και την εδαφική συνοχή. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση της ηγήτριας για την εξάλληψη της χρηματοδότησης για τα σύνορα ε, και την ασφάλεια με το επιχείρημα ότι αυτά καλύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα και ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Ταμείο Ασύλου ή Εσωτερικής Ασφάλειας. Αυτά τα ταμεία μπορεί να καλύπτουν σε έναν βαθμό αυτούς τους τομείς, ωστόσο κατευθύνονται κυρίως στα κράτη-μέλη της Ένωσης και όχι στις υποψήφιες χώρες. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν, ε, ωστόσο, όπως και η συγγήτρια, ε, σοβαρά εχέγγυα για την αποφυγή αλληλεπικάλυψης στη χρηματοδότηση, ώστε η ίδια δράση ποτέ να μην χρηματοδοτείται δύο φορές από δύο διαφορετικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, προσβλέπουμε και στην επικοδηματική συνεργασία με την συγγήτρια σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η Κομισιόν θέλει το λόγο, παρακαλώ. Μόνο αν έχετε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επισημάνω ότι είχα φύγει από την αίθουσα για να παρακολουθήσω την, το σεμινάριο για τα Δυτικά Βαλκάνια που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και εκεί γίνεται μια συζήτηση για τη μία απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι πολλές δράσεις που σχετίζονται με την ε, άμβλυνση της ακραίας φτώχειας δεν ε, χρηματοδοτούνται, δεν αξιοποιούνται τα κονδύλια για διάφορους λόγους και ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, το θέμα αυτό και από ακαδημαϊκής άποψης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει η βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα ε, χαρακτηριστικά. Διότι το πρόβλημα είναι ότι τους δίνουμε χρήματα, δεν τα αξιοποιούν και έτσι, το πρόβλημα, και, και έτσι τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Με τον διάλογο και μέσω της ε, χρήσης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ίσως θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε κάποιες δέσμες μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που ε, αντιμετωπίζουν. Εγώ θα μπορούσα να κάνω τέτοιε προτάσει για τη φτώχεια, για παράδειγμα, ή για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να αναλάβει κανεί για να ε, καταπολεμήσει το τράφικινγκ, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλα τα χρήματά μα να συνοδεύονται από αυτό που είπα, από συγκεκριμένε προτάσει για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ε, αξιοποιηθούν από τι υποψήφιε χώρε. Πρόεδρο, να ε, ξαναδώσω το λόγο στην Πόντιλ για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω, έχουμε εκπρόσωπο της Κομισιόν. Α, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώς ορίζει τη γνωματότηση της κυρίας Βαλέρο και κυρίως τη σημασία που βλέπουμε σε όλη την έκθεση για το μηχανισμό ως μακροπρόθεσμη επένδυση στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Σημειώνουμε ότι συζητάτε σε κάποιους τομείς ε, να δοθεί έμφαση κοινωνική συμπερίληψη, κοινωνική άμα, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, συνοχή. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η τομή προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πρόταση του κανονισμού μπορείτε να βρείτε κάποιου από αυτού του τομεί, οι οποίοι απαριθμούνται στι θεματικέ ενότητε, ε, στα Προσαρτήματα έχουμε λοιπόν τους ε, θεματικές ενότητες και επίσης κάποιους τομείς ε, σημασίας οι οποίοι είναι για παράδειγμα η διεθνής προσοχή και στο παράρτημα 2 στόχος D στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη θα βρείτε κάποιες υποθεματικές ενότητες οι οποίες ε, ακριβώς κινούνται στην κατεύθυνση της αύξησης της κοινωνικής συνοχής. Σημειώνουμε επίσης και συμφωνούμε για την ανάγκη να αποφύγουμε επικάλυψη οποιοδήποτε μέσων που σχετίζονται με την μετανάστευση. Από την άποψη αυτή, συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά στην προετοιμασία του Πουδουπού σε ένα σημείωμα για το πώς θα πρέπει να εναρμονιστεί τα εσωτερικά και εξωτερικά οικονομικά μέσα τα οποία έχουν να κάνουν με την μετανάστευση και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και αν θέλετε μπορούμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη δουλειά που κάνετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος, και να δώσουμε το λόγο στην Πόντιλ για να κλείσει. Να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο και προσβλέπω στις τροπολογίες. Θα τις κοιτάξω. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχόλιά σας. 3 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 5 το απόγευμα. Και μετά θα εξετάσουμε τις τροπολογίες φυσικά. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή είναι 10 Ιανουαρίου. Αυτό λέει το χρονοδιάγραμμα στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 28, λέει ο Πρόεδρος. Να περιμένουμε τον κύριο Νίτερ Μιούλερ για το 28, Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Okay, colleagues, I'm just advised that we pause. I'm sorry. Συνάδελφοι, δέκα λεπτά διάλειμμα. Μέχρι να εκτεφτάσει ο κύριος Νίντερ Μούλερ. Ζητώ συγγνώμη γιατί είχαμε πολλές τέτοιες ε, αναστατώσεις ε, σήμερα το πρωί. Γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες παράλληλες συνεδριάσεις. Mr. Niedermüller is on his way. Also, we, we, we're, we're running uh, ahead of schedule also. Και είμαστε και μπροστά από την ώρα μας. Θα ξεκινήσουμε σε 10 λεπτά 28. Dear colleagues, thank you for your patience. We can begin on point 28, which is the... Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τον, για το άσυλο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Νίντερμιουλερ για το θέμα αυτό. Κανονικά θα μιλούσαμε για σχέδιο έκθεσης, αλλά έπρεπε να ακολουθήσουμε μια κάπως διαφορετική διαδικασία όπου παρουσιάστηκε τροποποιημένη πρόταση κομισιών στους συνομαφέτες παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή μας είχε ήδη εκδώσει εντολή ε, το 2016 και παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις οι οποίες διεξήχθησαν το 2017. Ε, ο εισηγητής εκ μέρους του Κοινοβουλίου έχει ήδη αποστείλει επιστολές στην Κομισιόν και στην, Ευρω... και Αυστρική Προεδρία και τους επισημαίνει ότι ε, το Κοινοβούλιο εμένει στην ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί. Σήμερα το πρωί έγινε μια συνάντηση για το πώς θα προχωρήσουμε. Ο κύριος Νίντερ Μιούλερ θα μας ενημερώσει για τα όσα διαμήφθησαν εκεί. Πέτερ, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είπες, υπάρχει μακρά ε, προϊστορία σε αυτό το θέμα. Και όπως ανέφερες, είχαμε ήδη ε, καταλήξει σε προσωρινή συμφωνία πολιτικού χαρακτήρα με τη Μαλτέζικη Προεδρία τον Ιούνιο του 2017. Μετά, για πολύ καιρό δεν είχαμε κάποια εξέλιξη και το Σεπτέμβριο του 2018 η Κομισιόν υπέβαλε νέα πρόταση υπό την ίδια διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο ε, και αυτό για ε, πολύ σημαντικούς λόγους. Το να επανυποβάλλεται ε, νέα πρόταση υπό, την ίδια, υπό τον ίδιο αριθμό διαδικασίας μετά την ε, ε, αφού το Κοινοβούλιο έχει ήδη καταλήξει στην εντολή του. Για να μπορεί το Κοινοβούλιο λοιπόν να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση από την πλευρά Κομισιόν ε, χρειάστηκε να βασιστεί στους δικούς του εσωτερικούς κανόνες. Όπως υπόθηκε λοιπόν, είχαν ήδη τον Ιούνιο του 2017 οι συνομοθέτες καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία και ανεξαρτήτως ε, του γεγονός ότι το κείμενο είχε παραπεμφθεί σε τεχνικό επίπεδο. Ε, είχε υπάρξει συμφωνία ε, συμπεριλαμβανομένης και της αιτιολογικής έκθεσης σε αγγίλες. Και παρά όλα αυτά, παρόλα αυτά, η Κομισιόν επανέρχεται με νέα τροποποιημένη πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι η νέα πρόταση της Κομισιόν δεν βοηθά του συνομοθέτε όσον αφορά την έγκριση του, της νέας ενωσιακής νομικής πράξης υπό την τρέχουσα θητεία. Αντιθέτως, ε, πολλαπλασιάζει ε, τα εμπόδια, καθώς η πρόταση καθίσταται πιο εξαρτημένη από ε, άλλους φακέλους που υπερβαίνουν και τα όρια του κοινού συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου το σύστημα της Ευρωπαϊκή Ένωση για το άστιλα να γίνει λειτουργικό το, ε, το συντομότερο δυνατό, η συμφωνία που είχε επιτευχθεί υπό Μαλτέζικη Προεδρία είναι ο μόνος δρόμος και ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε επανεξέταση μόνο εκείνων των σημείων που είχαν μείνει σε αγγίλες σε εκείνη τη φάση και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για αυτά και μόνο τα θέματα για να καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Στο επεξηγηματικό τη σημείωμα, η Κομισιόν ισχυρίζεται ότι έχει λάβει υπόψη τη την συμφωνία εκείνη που είχε ε, συναυθεί. Αντιθέτως όμως στην πραγματικότητα οι τροπολογίες της αλλάζουν ακόμη και επί της ουσίας το κείμενο. Και ακόμη πιο σημαντικό, ε, θεωρώ ότι η τροποποιημένη πρόταση είναι ελλειπής. Αν γίνουν αποδεκτές οι προτινόμενες αλλαγές και ενσωματωθούν από τους συνομοθέτες, η Κομισιόν προβλέπει ήδη άλλα τμήματα της ε, ε, προσωρινής συμφωνίας να ξανανοιχτούν όπως είναι η τεχνική βοήθεια, η ανάπτυξη ομάδων ε, για το άσυλο και διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα. Θεωρώ ότι η τρυπωμένη αυτή πρόταση ε, μας θέτει σε κίνδυνο να ξανανοίξουμε τη συζήτηση επί ολόκληρου του κειμένου. Για τους ε, λόγους αυτούς οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί ε, μεγάλη ε, μεταστροφή όσον αφορά την εντολή και τη λειτουργία του οργανισμού. Δεδομένης όμως της ανάγκης και του επίγοντος χαρακτήρα που έχει ο συγκεκριμένος ε, οργανισμός και η θέσπιση του, θεωρώ ότι η κίνηση αυτή από την Κομισιόν θέτει σε κίνδυνο το, μέλλον του ίδιου του οργανισμού. Είχαμε καταλήξει σε πολιτικό συμβιβασμό μεταξύ των συνομοθετών και με εκπλήσει το γεγονός ότι η Κομισιόν επανέρχεται με νέα τροποποιημένη πρόταση. Θέλω να ε, υπενθυμίσω και να επαναλάβω ότι η προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί υπό Μαλτεζική Προεδρία είναι η μόνη βάση επί της οποίας μπορεί να γίνει συζήτηση επί των κομματιών του κειμένου που είχαν τεθεί τότε σε αγγίλες. Το κείμενο της ε, προσωρινής συμφωνίας ε, πρέπει να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση και όπως είπα το πρωί, ε, είπατε, ε, είχαμε και μια άτυπη συνάντηση με τον ε, Επίτροπο Αβραμόπουλο και την Αυστριακή Προεδρία και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να προβούμε σε κάποια, να επιτύχουμε κάποια λύση και να προβούμε σε κάποιες συντονισμένες κινήσεις. Ευχαριστώ Πίτερ, λέει ο Πρόεδρος, και για την ενημέρωση της Επιτροπής μας. Ας ακούσουμε τους κοιόδες. Κάλλος Κοέλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όταν συζητήσαμε την πρόταση της Κομισιόν πέρσι τον, τον Οκτώβριο, με είπα ότι εξ όσων γνωρίζω έχουμε συμφωνία στο τραπέζι. Εξ όσων γνώριζα ήταν το πρώτο θέμα στο οποίο είχε επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία ε, ήδη πριν από δύο χρόνια σχεδόν. Δεν γνωρίζουμε γιατί η Κομισιόν ε, επέλεξε να κινηθεί με τον τρόπο που κινήθηκε και επίσης ε, εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε ε, ποιε είναι οι πραγματικές επιθυμίες του Συμβουλίου. Ξέρω όμω για το τι χρειάζεται να γίνεται. Πρέπει να εγκριθεί ο νέο οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το άσυλο και αυτό πρέπει να γίνει πριν από τη λήξη τη θητεία μα. Θέλουμε να επιτύχουμε τον στόχο αυτό. Η κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο εισηγητής μας είναι σωστή και μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξή μας. Βάση τη συζήτηση για εμά δεν είναι η τροπολογία τη Κομισιόν, αλλά η προσωρινή συμφωνία. Και γι' αυτό θα υποστηρίξουμε τον εισηγητή για να ακολουθεί μια ταχεία διαδικασία. Καλό την Κομισιόν και την Προεδρία να επιδείξουν την ίδια προσήλωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό αυτός ο νέος οργανισμός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά και υποστηρίζουμε λοιπόν αυτή την έτοιμα ε, για καταπήγοντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κάρλος ή Σοφή. Υποστηρίζω το θέμα αυτό με όλη μου την καρδιά και θα ήθελα να τονίσω πόσο ενοχλήθηκα. Καταρχάς, το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται να την χρησιμοποιεί το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τις ε, επιστροφές ε, δεν χρειαζόταν. Ενώ το Συμβούλιο μπλοκάρει οποιαδήποτε πρόοδο για το άσυλο. Είναι πραγματικά επονίδιστο, ανεύθυνο. Κοιτάξτε, πού οδεύουμε. τέταρτος χειμώνα, όπου ο κόσμος ζει στην Ελλάδα, στι σκηνέ. Εγώ προτείνω να πάει το Συμβούλιο στην Ελλάδα να ζήσει στις σκηνές και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρει γρήγορα μια συμφωνία. Γιατί αποδεχόμαστε λοιπόν να μιλάμε για τέτοια ζητήματα. Για, νέα, για νέους φακέλους, τη στιγμή που το Συμβούλιο δεν δέχεται να σημειώσει πρόοδο στο άσυλο. Δεν θα έπρεπε καν να συμφωνήσουμε ως θεσμικό όργανο επί της αρχής. Ευχαριστώ, Σοφή το μπλοκάρισμα του πακέτου για το άσυλο είναι πραγματικά κάτι το εξοργιστικό. Σα ευχαριστώ. Ποιο άλλο ήθελε το λόγο. Πρωτού ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ράιν, μετά την ήπια εισαγωγή, Σα χειραγωγεί το Συμβούλιο. Πάτε το λόγο να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την προτεραιότητα που έδωσε στο θέμα αυτό και για την ταχύτητα προετοιμασία του σχεδίου έκθεση. Να ευχαριστήσουμε επίση τον κύριο Ντερμιούλερ για την ευκαιρία που έδωσε στον Επίτροπο Αβραμόπουλο να μιλήσει στον εισηγητή και στους κοιόδες σήμερα το πρωί και νομίζω ότι αυτό ήταν ε, πολύ επικοδομητικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στη συνεργασία και στην ε, συνομιλίες μεταξύ των συνομοθετών για να ενισχυθεί στην τρέχουσα θετία ο οργανισμός. Και χαίρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που άκουσε ότι ο εισηγητής συμφωνεί με το όραμα ενός ισχυρού οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το άσυλο σε πυλώνα του ασύλου και ως μία υποστήριξη για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές πιέσεις. Γι' αυτό λοιπόν το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτά τα πολύ στοχευμένα μέτρα για τον οργανισμό, προκειμένου ο οργανισμός να έχει σαφή νομική εντολή για να δώσει την ε, λειτουργική ενίσχυση που χρειάζονται τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να τονίσω ότι η συνάντηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ παρουσιάστηκε η έκθεση αυτή. Η πρόταση λοιπόν αυτή, η τροποποιημένη αυτή πρόταση δεν ε, σκοπεύει να ανοίξει πάλι την ουσία της πολιτικής συμφωνίας που πετύχαν οι συνομοθέτες πέρσι. Γίνεται απόλυτα σεβαστή αυτή η ενδιάμεση συμφωνία. Αυτό που θέλει να κάνει η νέα πρόταση είναι να αναπτύξει αυτή την προσωρινή συμφωνία και να λάβει υπόψη τις εμπειρίες που είχαμε εν τω μεταξύ. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Ιταλία οι εμπειρίες αυτές καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα παραπάνω τη λειτουργία των συστημάτων που παρέχει ο οργανισμός προς τα κράτη-μέλη. Και για το λόγο λοιπόν αυτό ελπίζουμε το, συμβουλίο, το Κοινοβουλίο συγγνώμη, να συμφωνήσει με αυτές τις περιορισμένες αλλαγές οι οποίες βγάζουν νόημα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ε, αναφορές και τις επικαλύψεις με άλλα εργαλεία για το άσυλο που ανέφερε ο εισηγητής πολλά εξ αυτών είναι σε αγγίλες στην παρούσα φάση. Όλα αυτά μπορούν να επιληθούν γρήγορα σε τεχνικό επίπεδο. Αν χρειαστεί και με αναφορά στα εφιστάμενα μέσα, δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την ταχεία έγκριση του κειμένου. Προσβλέπουμε λοιπόν στην έναρξη των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε στο τεχνικό επίπεδο οποιαδήποτε ερώτημα ενδεχομένω έχουν τα μέλη. Πρόεδρος, έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι καλύτερα θα κάνουμε να τα συζητήσουμε κάτι Να Πίτερ, θέλεις να πάρεις το λόγο. Θέλει να πάρεις το λόγο. Όπως είπατε δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Έγινε αυτή η συνάντηση σήμερα το πρωί και συμφωνώ με την, Προεδρία, με την Επιτροπή. Ήταν επικοδομητική συνάντηση και ότι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φυσικά βλέπουμε τις ε, διάφορες και τις δυσκολίες της διαπραγματεύσεις αυτές, αλλά το Κοινοβούλιο πάντα προσπαθεί να επιτύξει η διάθεση. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. I'm having a meeting with the rapporteurs of... Θα συναντήσουμε τον εισηγητή, τους εισηγητές μάλλον από όλα τα τμήματα του πακέτου για το άσυλο. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την συνολική μας στρατηγική όπως είπε και η Σοφή. Έχουμε αντίληψη της κατάστασης. Ευχαριστούμε, Πίτερ. Ευχαριστώ και τους κοιότης. Προθεσμία για τα τροπολογιών. Είναι το Δεκέμβριο. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε, Πίτερ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 29. Okay. So, colleagues, this is the... Συνάδελφοι, είναι το τελευταίο σημείο για σήμερα, το πρωί. Κατάσταση στη Λιβύη και στην περιοχή έρευνας και διάσωσης. Γιατί το έχουμε αυτό στην ημερήσια διάταξη σήμερα, διότι αυτό το θέμα πανελειμμένα ήταν στην ημερήσια μας διάταξη. Στις 10 Οκτωβρίου έγινε συζήτηση με την UNHCR, την IOM και σε σχέση με τις πλατφόρμες αποβίβασης στην Μεσόγειο και ευρύτερα την κατάσταση. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε συνέχεια με μια σύντομη παρουσίαση. Ζητήσαμε δε μια γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία όσον αφορά την νομιμότητα των πλατφορμών αποβίβασης. Όλοι όσοι ήμασταν σε εκείνη τη συνεδρία ήταν αρκετά σημαντικοί και ευαίσθητοι. Ε, ε, οι συνάδελφοι θα έχετε δει τις διάφορες ε, αναφορές του τύπου. Κάναμε και συζήτηση με τους δημοσιογράφους που συνέταξαν αυτές τις εκθέσεις. Οπότε ξαναβλέπουμε αυτό το θέμα, του πού βρισκόμαστε ε, σε σχέση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου να ξανασυζητήσουμε και να ξαναεστιάσουμε ως Επιτροπή στο θέμα της έρευνας και της ε, διάσωσης εν γέννη, ε, τα κέντρα αποβίβασης, ε, τις πλατφόρμες αποβίβασης, τις συνέπειες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δεδομένης της πολύ ασταθούς κατάστασης στη Λιβύη. Ζητήσαμε από την Κομισιόν να μας μιλήσει για το θέμα που έθεσε η κυρία Βερζιά για την κατάσταση των προσφύγων για τους οποίους η προθεσμία εξέβνευσε τον Οκτώβριο δεν έχει απαντηθεί και γι' αυτό ζητήσαμε να μπει στην ατζέντα της Λιβύης για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και λόγω του εξαιρετικά δύσκολου πλαισίου και της κατάστασης και των ανησυχιών που έχουμε θα έχετε δει πως επιδεινώνεται η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση της ασφάλειας ε, στην χώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε την κατάσταση. Καλέσαμε διάφορους ομιλητές που θα πάρουν το λόγο. Ένας, δύο, ένας, δύο από τους ομιλητές μας δεν έχουν φτάσει ακόμα. Και επειδή όλοι ήσασταν πολύ υπομονετικοί σήμερα το πρωί, όπου είχαμε ένα σωρό ζητήματα με τους συναδέλφους που έπρεπε να είναι σε άλλες επιτροπές και τα λοιπά, λόγω αυτού θα ήθελα να προτείνω να ξεκινήσουμε με τους συνάδελφους ομιλητές που είναι παρόντες ήδη και μετά να προχωρήσουμε με τη συζήτησή μας. Αν συμφωνείτε όλοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την νομική υπηρεσία. Να θυμίσω ότι ζητήσαμε αυτή την γνωμοδότηση όσον αφορά τις περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβαση. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο ξερός αυτό ο τίτλο, αλλά πάει στην καρδιά των συμπερασμάτων, των πορισμάτων μάλλον του Συμβουλίου. Δεν έχει λυθεί κατά το πρόβλημα παρά τα όσα κάνει το Συμβούλιο. Η γνωμοδότηση αυτή λοιπόν θεωρείται εμπιστευτικού χαρακτήρα. Πού είναι ο Ντάνιελ? Ο Ντάνιελ έχει το λόγο να μας την παρουσιάσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή έχει συνταχθεί στα αγγλικά, παρόλα αυτά εγώ θα μιλήσω στα γαλλικά. Όντω η Επιτροπή σα ζήτησε την ε, γνώμη της νομικής υπηρεσίας όσον αφορά τη συμβατότητα των πλατφορμών, ε, περιφερειακών πλατφορμών αποβίβασης και των ελεγχόμενων κέντρων όπως προτείνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28 Ιουνίου 2018. Η δυσκολία αυτού του εγχειρήματο έγκυται στο ότι η έννοια που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, οι έννοιες μάλλον αυτές δεν ήταν πολύ αναπτυγμένες και κάλυπταν πραγματικότητες με τις οποίες μάλλον για τις οποίες ήταν δύσκολο να εκφραστούμε πολύ συγκεκριμένα, επειδή δεν γνωρίζαμε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσαν αυτές οι δομές λεπτομερώς η διαφορά ανάμεσα στις δύο έννοιες, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις πλατφόρμες αποβίβασης και το και κέντρου, ελεγχόμενων κέντρων δεν υπήρχε εξαφή διαχωρισμό. Αυτές οι πλατφόρμες, από ό,τι φαινόταν, στόχο είχαν να εγκατασταθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ελεγχόμενα κέντρα θα ε, έπρεπε να λειτουργήσουν στην επικράτεια τη ένωση. Αυτό κατέληγε κανείς διαβάζοντα τα απορρίμματα του Συμβουλίου. Όμω, η δυνατότητα για πλατφόρμες αποβίβαση εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον εντό τη Ένωση, επίσης είχε ε, αναφερθεί και μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εφόσον έχουμε πλατφόρμες αποβίβασης εντός της Ένωσης, δεν είναι εύκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα στις δύο έννοιες, γιατί οι στόχοι είναι παρόμοιοι, αρκετά παρόμοιοι, διότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πρόκειται για ε, μια γρήγορη ε, διάκριση ανάμεσα στους μετανάστες, ώστε να αποφασίσουμε ποιοι από αυτούς δικαιούνται διεθνή προστασία και ποιοι όχι. Εν πάση περιπτώσει, τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη όταν θέλει να εκτιμήσει την νομιμότητα τέτοιων δομών είναι η εγκατάστασή τους ή όχι στην επικράτεια της Ένωσης. Θα εξετάσουμε λοιπόν πρώτα τις δομές, όποιο και θα είναι το όνομα που θα λάβουν τελικά, που θα εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται να είναι δύσκολο να εντοπιστούν εμπόδια στην εγκατάσταση αυτή. δεδομένου του στόχου που τους ανατίθεται και που είναι συμβατός με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ασύλου, Τέτοιες δομές μπορούν λοιπόν ε, ε, καταρχήν νόμιμα να εγκατασταθούν στην επικράτεια της Ένωσης για να υποδεχτούν τους μετανάστες, είτε αυτοί ε, έχουν σωθεί στην επικράτεια της Ένωσης, δηλαδή και στα ύδατα των εγχώρια ύδατα των κρατών μελών, είτε στην στεριά. Σε αυτό το στάδιο δεν διευκρινίζεται τίποτα όσον αφορά αυτούς τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των δομών. Και άρα η διτομική υπηρεσία δεν μπορεί να εκτιμήσει πολύ συγκεκριμένα ποια θα είναι η πραγματικότητα αυτή ακριβώς. Πάντως οι δομές αυτές θα υπόκειται άμεσα και εξ ολοκλήρου στο δίκαιο του ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, ως προς αυτό Η γνωμοδότηση που σας δίνουμε αφορά μόνο την ε, ακαιρεότητα των μεταναστών γιατί η ιδέα και μόνο ε, θέτει αυτό το ζήτημα. Ότι δηλαδή ο όρος του ελεγχόμενου κέντρου θεωρείται ε, ότι παραπέμπει σε κλειστά κέντρα κράτησης. Ως προς αυτό η οδηγία 2013-33 για τις συνθήκες υποδοχής των ετούντων άσυλο διευκρινίζει και προβλέπει ότι οι ετούντες άσυλο χαίρουν εν γέννη της ελευθερίας κίνησης στην επικράτεια των κρατών ε, που τους υποδέχονται. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι μπορεί να επιβληθούν ε, περιορισμοί σε αυτή την ελευθερία κίνησης, κυκλοφορίας, χωρίς ε, να διευκρινίζονται ή να προκαθορίζονται συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Απλά πρέπει αυτοί οι περιορισμοί να μην απομονώνουν τελείως, να μην επηρεάζουν μάλλον την σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και να επιτρέπουν στον δικαιούχο να μπορεί να ε, εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα και τις εγγυήσεις που του προσφέρει η ίδια η οδηγία αυτή. Εξάλλου, τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν στους ετούντες άσυλο μια, κάποιο χώρο ε, διαμονής μέσω μιας ε, γενικής απόφασης και άρα, επί της αρχής, η ιδέα του να προβλεφθούν ελεγχόμενα κέντρα όπου οι μετανάστες συγκεντρώνονται μπορεί να είναι συμβατή με τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης για αυτά τα θέματα. Και πάλι, βέβαια, υπό την επιφύλαξη του τι ακριβώς θα προβλέψει το κείμενο το οποίο θα θεσπίσει και θα δημιουργήσει αυτά τα ε, κέντρα. Περιορισμός της κυκλοφορίας μέσα σε αυτά τα κέντρα επίσης θίγει, ε, ακόμα κι αν ε, να επαναλάβω ότι ήταν, ε, δεν, δεν κατέστη δυνατό να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η κράτηση των ετούντων άσυλο πρέπει να θεωρείται ως εξαίρεση που θα πρέπει να προβλέπεται από το νόμο και που θα πρέπει να υπόκειται στην αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Ένα μέτρο κράτησης ε, δεν μπορεί να εφαρμόζεται γενικά και αόριστα, αλλά κατόπιν ατομικής εξέτασης ε, μεμονωμένων περιστάσεων. και θα μπορεί να εφαρμόζεται μέσα στο πλαίσιο και εφόσον τηρούνται ε, κριτήρια συγκεκριμένα τα οποία θα ορίζονται από το νομικό κείμενο. Αυτά μπορούμε να πούμε σε αυτό το στάδιο για τέτοιου είδους δομές στην επικράτεια της Ένωσης. Για τους ανθρώπους που και για την ε, κέντρα αποβίβασης, μάλλον πλατφόρμες αποβίβασης που θα βρίσκονται εκτός της Ένωσης. Η νομική αξιολόγηση που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το στάδιο είναι πιο περίπλοκη και εξαρτάται από το τόπο διάσωσης των μεταναστών που θα οδηγηθούν σε αυτές τις δομές. Αν αυτοί οι μετανάστες έχουν σωθεί, διασωθεί στη χώρια ήδη μιας χώρας εκτός Ένωσης, οι μετανάστες αυτοί δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία κάποιου κράτους μέλους της Ένωσης και άρα βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του ευρωπαϊκού ε, δικαίου περί ασύλου ωστόσο καλύπτονται από το δίκαιο του, της τρίτης χώρας που θα τους υποδεχτεί και από τις διεθνείς συμβάσεις. Δηλαδή, η Σύμβαση της Γενέβης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων από τη στιγμή που ε, το, κράτος, το εν λόγω κράτος έχει υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Ωστόσο, εάν η Ένωση ε, προβεί σε άτυπη ή τυπική δέσμευση για να σχεδιάσει και να λειτουργήσει τέτοιου είδους πλατφόρμες εκτός Ένωσης, αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να σέβονται τις εγγύσεις που προσφέρει η Σύμβαση της Γενέβης και κυρίως την αρχή της μη απόθεσης που επιτρέπει στην δημιουργία τέτοιων πλατφορμών μάλλον απαγορεύει την δημιουργία τέτοιων πλατοσφορμών σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς. Όσον αφορά τους ε, μετανάστες που διασώζονται στην ανοιχτή θάλασσα, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι καλύπτονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι δεν βρίσκονται στην επικράτεια κάποιου κράτους μέλους δεν σώζονται στην επικράτεια κάποιου μέλου. Ακόμα κι αν διασωδούν από κάποιο πλοίο που φέρει τη σημαία κράτου μέλου, εκτός από συγκεκριμένε περιστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη γνωμοδότηση. Γιατί εν γέννη είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι ένα σκάφος που φέρει τη σημαία ενός κράτου μέλους αποτελεί προέκταση του ίδιου του κράτου μέλους και τη δικαιοδοσία αυτού. Άρα λοιπόν ο μετανάστης που διασώζεται στην ανοιχτή θάλασσα μπορεί να θεωρηθεί όπως και οι υπόλοιποι μετανάστες που διασώζονται εκτός της επικράτειας της Ένωσης. μόνο για τους μετανάστες που διασώζονται στα ύδατα μιας χώρας μέλους της Ένωσης, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, στα ευρωπαϊκά χώρια ύδατα, αυτοί δεν μπορούν να σταλούν εκτός της Ένωσης χωρίς να έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Ασύλου και χωρίς να έχει διεκπαιρεωθεί και εξεταστεί πλήρωση το αίτημα ασύλου τους. Κάτι τέτοιο θα θεωρείται απόθεση που απαγορεύεται κάθετα τόσο από τη Σύμβαση της Γενέβης όσο και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η προστασία αυτή λοιπόν δεν μπορεί να δοθεί στους μετανάστες που θα μεταφερθούν στη κέντρα εκτός ε, της Ένωσης και δεν μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις σε κέντρα τα οποία θα βρίσκονται, όπως σας είπα, εκτός της Ένωσης. Δεν βλέπουμε λοιπόν πώς οι μετανάστες που μπορεί να διασωθούν στη χώρα ήδη ενός κράτους μέλους μπορούν να στέλνονται σε πλατφόρμες ε, κοινού δικαίου εκτός της Ένωσης. Αυτά είναι, αυτό είναι το ζουμί αυτής της νομοδότησης που όπως σας είπα είναι περιορισμένη διότι τελικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοούσε το Συμβούλιο για τις συγκεκριμένες δομές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για κάθε σας ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν θαραλέα η προσπάθειά σας με τα, όσα έγιναν από τον Ιούνιο από το Συμβούλιο, από την Κομισιόν, τα έγγραφα που εκδόθηκαν. Ίσως θα μπορούσε η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Πίεση της Εξωτερικής Δράσης να μας πούν κάποια στοιχεία σε σχέση με το που βρισκόμαστε όσον αφορά αυτά τα δύο έγγραμμα. Παρ' όλα αυτά, ήταν θαραλέα η, προσπάθειες, η προσπάθειά σας για να δούμε, να δείτε πού βρισκόμαστε. Οι πλατφόρμες αποβίβασης μπορούν να βρίσκονται και εντός και εκτός. Δηλαδή μπορεί να είναι τα πάντα και τίποτα. Είναι σαν ε, έργο του Κάφκα. το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούσατε να κάνετε είναι αυτή η αναφορά σας στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ε, το είπατε ε, έξι φορές ότι το ενωσιακό δίκαιο ισχύει στην επικράτεια και τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να φανώ ε, Δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο από τον Ιούνιο καθόλου. Θετικό είναι το γεγονός ε, πάντω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατέληξε σε μια νομική γνωμοδότηση, η νομική του υπηρεσία, για την ανάγκη εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε περίπτωση που είχε κάποιος άλλε προθέσεις ή άλλε ιδέες. Συζητάμε λοιπόν με τον IOM, με την ύπατη αρμοστία, αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Οπότε νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε και στο, στην ερώτηση της κυρίας Βερζιά. Για εκείνους που κατέφτασαν αργοπορημένοι, να εξηγήσω τι κάνουμε. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία ε, και να ενημερωθούμε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη. Επόμενη κίνηση θα είναι η ερώτηση προς την Κομισιόν σχετικά με τους ε, πρόσφυγες που κρατούνται ε, στην Λιβύη. Νομίζω ότι μπορούμε να απευθύνουμε το ερώτημα αυτό στην Κομισιόν. Εντάξει, η κυρία Βεζιά δεν είναι εδώ. Η κυρία Σπινέλη όμως θέλει να αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν για να μας απαντήσει. Μπάρμπαρα, αν μπορείς, σε παρακαλώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ εδώ την κυρία Βερζιά που δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρούσα σε αυτή μας τη συνεδρίαση. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 υπέβαλε γραπτή ερώτηση κατά προτεραιότητα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία είχαν συνυπογράψει περίπου 20 βουλευτέ, ευρωβουλευτές από διάφορες ομάδες αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει απάντηση από την Κομισιόν παρά στον πήγουσα ε, ανθρωπιστική κατάσταση που αφορά ε, την ολοένα και επιδεινούμενη κατάσταση των προσφύγων που κρατούνται στη Λιβύη. Υπάρχουν περίπου 8.000 μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί από τη διεθνή κοινότητα και οι οποίοι χρειάζονται κατεπηγόντως προστασία, τρόφιμα και ιατρική φροντίδα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες αναφορές που επιβεβαιώνουν πως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση ούτε στην, σε τροφή ούτε στο νερό. Και κατά συνέπεια επικρατεί η κατάσταση λοιμού και εμπορίας ανθρώπων. Ο ύπατος εκπρόσωπος ε, του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Ε, πρότεινε και την ύπαρξη μιας κοινή θέσης για την προστασία των μεταναστών που διασώζονται στη θάλασσα και οι οποίοι δεν θα πρέπει να ε, στέλνονται στη Λιβύη. Ποιες είναι οι Ποια είναι τα βήματα που σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για να απελευθερώσει τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες που είναι φυλακισμένοι στην Τρίπολη. Ε, δεύτερη ερώτηση είναι η Κομισιόν έχει την πρόθεση ή όχι να αναστείλει την ενίσχυση που έχει ε, προβλέψει για την ε, ακτοφυλακή της Λιβύης, ώστε οι άνθρωποι που διασώζονται στη θάλασσα να μην παραπατρίζονται σε χώρους όπου η ζωή τους τίθεται άμεσα σε κίνδυνο. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε Μπάρμπαρα. Από την Γενική Διεύθυνση ε, Εσωτερικών Υποθέσεων έχουμε μαζί μας τον εμπειρογνώμονα της Κομισιόν για τη Λιβύη. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Πρωτού το ξεχάσω όμως θέλω να πω το εξή. Ε, να χρησιμοποιείτε ε, τον, όρο ελεγχόμενα κέντρα. Δεν καταλαβαίνετε ποιο είναι το ιστορικό φορτίο τέτοιων, όρων. Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι θα βάζετε τους ανθρώπους σε ελεγχόμενα κέντρα. Ούτε, ούτε καν το πιάνετε, δεν το καταλαβαίνετε. από άποψη ουσίας το πράγμα είναι ήδη αρκετά κακό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε και έναν τόσο φορτισμένο όρο. Καταλαβαίνετε ότι ε, πλήττεται το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί και να μην εκφράζω κανένα παρά μόνο τον εαυτό μου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάτι τελείως διαφορετικό ιστορικά. Πέρα από αυτά, πείτε μας και πού βρισκόμαστε ακριβώς, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σχέση με αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι από πλευρά Κομισιόν το κοινοβουλευτικό ερώτημα βρίσκεται σε φάση ε, ε, σύνταξης της απάντησης, η οποία θα αποσταλεί σύντομα στο Κοινοβούλιο. Να σας δώσω και εγώ κάποιες ε, κάποια ενημέρωση σε σχέση με, τις... με τα κέντρα και την περιοχή έρευνας και διάστασης που συζητάμε και σήμερα. Να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Συνολικός αριθμός αφήξεων στις 21 Νοεμβρίου ήταν γύρω στις 22.000 άνθρωποι, δηλαδή 80% λιγότερο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017. Τώρα να αναφερθώ λίγο στο πλαίσιο Η περιοχή έρευνα και διάσωση είναι μια περιοχή στην οποία ισχύει το διεθνέ δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα ούτε να συντονίζει ε, αυτές τις ε, δραστηριότητες ούτε και να προσδιορίζει ποιοι θα είναι οι χώροι αποβίβαση. Βεβαίω, αυτό δεν σημαίνει ότι μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Συνεχίζουμε ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μα να παρέχουμε συνδρομή στις τεχνικές επιχειρήσει. Ε, για τα κράτη-μέλη, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε και να διευκολύνουμε την επίτευξη βιώσιμων λύσεων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνετε υπόψη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ικανότητες ε, και ο συντονισμός γύρω από την έρευνα και τη διάσταση, καθώς και η αποτελεσματικότητα ε, στον τομέα αυτό, έχουν αυξηθεί σημαντικότατα χάρη στις παράκτιες χώρες, στο συντονισμό των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίω του Frontex, καθώς και τις κοινέ ε, ναυτικές επιχειρήσεις, όπως ήταν η επιχείρηση Σοφία και βεβαίως την αξιέπαινη συμβολή των ε, ΜΚΟ. Να αναφερθώ εδώ και στην κοινή επιχείρηση της οποίας ε, ηγήθηκε η Frontex για να καταλάβουμε ποιες είναι οι διατάξεις που ε, υπάρχουν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της επιχείρησης για την έρευνα και διάσωση. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ε, η αναλογία ε, και η ο στόχος της επιχείρησης είχε και την, ε, τη διάσταση της έρευνας και της διάσωσης. Ωστόσο, οι ερμοδιότητες ε, του Frontex ε, περιορίζονται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό. Κάθε ένας έχει βεβαίως νομικό και ηθικό καθήκον να βοηθά εκείνους που πνίγονται στη θάλασσα Ωστόσο, ε, θα πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Αυτό ήταν και το βασικό καθήκον, η βασική υποχρέωση ε, και στόχος της ε, επιχείρησης της οποίας ηγήθηκε ο Frontex. Το 2018 ο οργανισμός συμμετείχε σε 86 τέτοιες δράσεις διάσωσης, διασώζοντας περίπου 4.000 900 μετανάστες. Αυτά όσον αφορά την εμπλοκή του οργανισμού στις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης. Όσον αφορά τη λιβική ακτοφυλακή και τη συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, γνωρίζουμε όλοι ότι η ακτοφυλακή της ε, Λιβύης έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως ε, νόμιμη δομή αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων. Πολλά μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να υποστηριχθεί η ακτοφυλακή της Λίβυης και βάσει των ε, πληροφοριών που έχουμε από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης το 2018 η ακτοφυλακή της Λιβύης συνέβαλε στην διάσωση πάνω από 40.000 ε, μεταναστών που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα. Από αυτή την άποψη θέλω επίσης να επισημάνω και την ε, συμβολή και τη συνδρομή του Frontex ε, όσον αφορά την, κατάρτιση της ακτοφυλακής της ε, ε, Λιβύης. Μέσω μεταξύ άλλων της επιχείρησης ε, Σοφία παρέχοντας ε, συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης ε, στο προσωπικό της ακτοφυλακή τη ε, Λιβύης. Επιβεβαιώνω ότι στι προγραμματιζόμενες εκπαιδεύσει υπάρχει πάντοτε και ένα συγκεκριμένο μάθημα, ένα συγκεκριμένο κύκλο που αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελευταίο σημείο που έχει τεθεί τα τελευταία πολλά χρόνια σχετίζεται με τις ε, δραστηριότητες διάσωσης που διεξάγουν οι λιβικές αρχές. Οι αρχές αυτές έχουν ενημερώσει τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οργανισμό του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα και που δεσμεύεται από τη Σύμβαση του Αμβούργου, τη Σύμβαση για την ε, ε, Ασφάλεια της Ζωής στη θάλασσα, οι λιβικές αρχές λοιπόν έχουν ενημερώσει τον ε, ε, IOM για την περιοχή έρευνας και διάσωσης που είναι μια μονομερής ενέργεια όπως προβλέπεται άλλωστε γιατί έχει τις σχετικές αρμοδιότητες η Λιβύη και βεβαίως αντίστοιχα οι αρχές της. Προσδιορίσαν λοιπόν οι λιβικές αρχές ακριβώς τα γεωγραφικά όρια αυτής της περιοχής και την ε, εθνική αρμόδια ε, αρχή που έχει ορίσει η χώρα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι ως αποτέλεσμα της διακήρυξης αυτής της περιοχής οι λιβικές αρχές έχουν στείλει και ένα σχέδιο συμφωνίας ε, στις γειτονικές χώρες, Αίγυπτο, την Ισία και Ιταλία. Δεν απεστάλλει όμως το σχέδιο συμφωνίας αυτό στην Μάλτα, διότι πιστεύουν ότι μια διμερή συμφωνία έρευνας και διάσωσης με τη Μάλτα που, που έχει υπογραφεί με τη Μάλτα από το 2009 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Αυτή είναι η κατάσταση. Να... Δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω για την κατάρτιση και τη συνεργασία που έχουμε με τι λιβικές αρχές, γιατί είναι εδώ και ο εκπρόσωπο ο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση που θα σας τα πει. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ σοβαρές και αυστηρές διαδικασίες επιλογής προσωπικού κάθε φορά που θα υποδεχόμαστε εδώ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπαιδευόμενους ε, μέλη και στελέχη των λιβικών αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και προτείνω τώρα να ακούσουμε τον κύριο Πικέ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον κύριο Κασέντα από τον IOM και τον Δόκτωρ να αλλάξει. Αν θα μπορούσατε παρακαλώ όλοι σας να είσαστε σχετικά σύντομοι. Η Σοφή, μην Ακούσαμε πολλές ε, τεχνογραφικές εξηγήσει. Δεν πήραμε απάντηση στην ερώτησή μας. Είναι απλή ερώτηση μας. Τι κάνετε για να εγκαινώσετε τον κόσμο και για να εξασφαλίσετε ότι δεν ε, είναι σε ένα σημείο όπου οι ζωές τους είναι σε κίνδυνο. Ναι, και εγώ αυτό θέλω. Θέλω λίγο πιο πολύ χρόνο για τη ε, συζήτηση. Ναι, μα θα απαντήσετε την ερώτηση. Υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν απάντησε ο Πρόεδρος. Αν σας ακούσουμε όλους σας, ακόμα και αν είστε λίγο σύντομοι μάλλον, Τι προτείνω. Να μην ακούσουμε ε, παρουσιάσεις μεγάλες παρουσιάσεις. Αλλά μια σύντομη παρέμβαση και εξήγηση των σημείων κλειδί. Για να απαντήσουμε κάποιες βασικές ερωτήσεις. Είδαμε τι συνέβη πρόσφατα. Πείτε μας τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να ξέρουμε. όχι μεγάλες παρουσιάσεις, αλλά μιλήστε μας 4-5 λεπτά και πείτε μας τα σημεία κλειδί. Τα γνωρίζετε τα θέματα σας, άλλωστε καλά όλοι σας. Και μετά να ακούσουμε το καταιγισμό ερωτήσεων που περιμένω, γιατί και εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Ο κύριος Πικέ. Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα βασικά σημεία που έχουν αναφέρει είναι το εξή, ότι καταρχάς αυτή η συζήτηση προχωράει στο Συμβούλιο. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής. Δεύτερον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στα διάφορα θέματα και στους διάφορους φακέλους των τελευταίων χρόνων και τόνισα ότι Ό,τι και να γίνει για την ε, συζήτηση για την αποβίβαση θα πρέπει για τα κέντρα αποβίβασης συνεργαζόμαστε σε πολλά ζητήματα για την ενίσχυση των, ε, της ασφάλειας συνόρων για να υπάρξουν σχετικοί θεσμικοί φορείς και κατάρτιση αυτών. Ξέρετε πως έχει αστάθεια στη Λιβύη. Είναι δύσκολο. Ξέρετε τι προβλήματα έχουμε στο Νότο. Υπάρχει μια κατάσταση ατιμορρησίας και έλλειψης κυβέρνησης. Κατά δεύτερον, ακούμε ότι έχουν ξεμείνει μετανάστες ε, και πρόσφυγες στη Λιβύη και άτομα στους καταβλισμούς κρατήσεις. Παράχουμε λοιπόν βοήθεια μέσω της συνεργασίας με ΜΚΟ και με ανθρωπιστικές οργανώσεις για την ε, επίσης ε, δημιουργία υγειονομικής ε, περίθαλψης, εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης στο βαθμό του δυνατού σε αυτές τις καταβλισμούς. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις αρχές της Λιβύης όπως μπορούμε και όταν έρχονται αντιπροσωπείες τους εδώ στις Βρυξέλλες και όταν εμείς μεταβαίνουμε εκεί, όπως συμβαίνει τώρα. Και έχουμε τέλος επαναπατρίσει σε ανθρωπιστική εθελούσια βάση 34.000 ανθρώπους, άτομα που μας ανησυχούν στη χώρα προέλευσής τους και τους έχουμε διασώσει από τις φρικτές συνθήκες που έχουν ρίσει στα κέντρα κρατήσει. Τρίτο επίπεδο, καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος τράφικες ε, ανθρώπων ε, είδαμε με την επιχείρηση Σοφία ότι έχουν έξι υποτεροριστεί 230 σκάφη διακινητών και το πρόβλημα αυτό το καταπολεμούμε και μέσω ε, ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Europol, Frontex και Σοφία. Πρόσφατα επιβληθήκαν κυρώσεις για εγκληματίες που κάνουν εμπορία ανθρώπινων ανθρώπων. Υπάρχει αυτό το εργαλείο επιβολής κυρώσεων στο Σοφία, να προσθέσω. Ότι έχουμε την καταπολέμηση των διακινητών, αλλά έχουμε και τη διάσωση των ανθρώπων από τη θάλασσα. 3.000 άτομα έχουν με τον τρόπο αυτό. Τέλος το πρόβλημα μετανάστευσης στη Λιβύη θα επιληθεί βιώσιμα μόνο αν υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνική κατάσταση μέσα στη Λιβύη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό. Απασχολεί ιδιαίτερα και την ε, είπατε εκπρόσωπο. Ήταν στο Παλέρμο πριν από μια δεκαετία ημέρε και δεσμευτήκε πλήρω για τη χρήση και την ε, χορηγήση κάθε δυνατή υποστηρίξη από πλευρά τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προ του Οργανισμού ε, των Ηνωμένων Εθνών. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. και τώρα α περάσουμε στην, στον Πατρί Ξέντα, εμπειρογνώμονα από την Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευση. Σα ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα μαζί μα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνεται να απευθυνθούμε στην Επιτροπή σας. Θέλω να κάνω τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις εισαγωγικά ε, συγκεκριμένα για τη Λιβύη και την κατάσταση των μεταναστών. Η σταθερότητα της χώρας είναι αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο. Ξέρετε ότι πέρα από τους μετανάστες υπάρχει μια φρικτή ανθρωπιστική κατάσταση ε, εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, υπάρχουν εσωτερικώς εκτοπισμένοι στη χώρα που και αυτά θα πρέπει να μην ξεχνιούνται στη συζήτηση. Να σας δώσω μια αίσθηση για τον αντίκτυπο της κατάστασης στην ασφάλεια, στις ε, δράσεις μας. Ε, έχουμε βοηθηθεί από τα 253 μέλη του προσωπικού μας που εργάζονται σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Έχουμε 9 διεθνείς εργαζόμενους που έχουν ε, αναπτυχθεί, που εργάζονται επί τόπου. Δυστυχώς οι κανόνες δεν μας επιτρέπουν ε, να διευρύνουμε τον αριθμό των εργαζομένων. Ελπίζουμε όμως ότι αυτό θα καταστεί εφικτό από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Οι επιχειρήσεις μας ε, έχουν ως έδρα τους και βάση τους στην Τρίπολη. Προσπαθούμε όμως να ανοίξουμε τις δράσεις μας και στην, στο, στην και σε άλλες χώρες, αλλά ξέρετε ότι και σε άλλες πόλεις αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Αυτό θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής της διεθνούς κοινότητας και των δράσεων της. Όσον αφορά τους ε, μετανάστες που επιστρέφονται από την ακτοφυλακή της Λιβύης, ε, υπήρχαν κάποιες επιστροφές που έγιναν αυτό το μήνα, περίπου 500 άνθρωποι. Συνολικά από τις αρχές του χρόνου μιλάμε για περίπου 15.000 ανθρώπους που διασώθηκαν από την ακτοφυλακή της Λιβύης και αυτό ε, πρέπει να το συγκρίνει κανείς με τις αφήξεις στην Ιταλία ε, γύρω στις 22.000 φέτος ρεκόρ χαμηλών αφήξεων για τα τελευταία χρόνια 1268 νεκροί από την αρχή του χρόνου. Αυτό έγινε και στην Μισράτα, στο πλοίο, όπου μετανάστες αρνήθηκαν να αποβιβαστούν. Από διάφορες χώρες κατάγονταν, κάποιοι μάλιστα ακόμη και από τον Μπαγκλαντές. Ε, πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης. Ε, επίσης, Προσπαθούμε να αναπτύξουμε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στην έρημο με την υποστήριξη των λιβικών αρχών προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στις δραστηριότητες μας. Ε, ξέρετε ότι ήδη δραστηριοποιούμαστε στα σύνορα με την Ιγυρία αλλά και η κατάσταση εκεί ε, επιδεινώνεται και δυσκολεύεται λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Οι μετανάστες ε, ε, ε, επιστρέφονται σε κέντρα κράτησης ένα, μια επιδίωξη, ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε αναπτύξει, επισημάνει και εμείς και η Πατεαρμοστία. 26 τέτοια υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα και εκεί φιλοξενούνται λίγο παραπάνω από 5.000 άνθρωποι. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 όταν και ξεκινήσαμε μια μεγάλη κλίμακα επιχείρηση ε, εκένωσης. 17.000 άνθρωποι κρατούνταν τότε, είναι πλέον 5.000 με κάποιες διακυμάνσεις ανάλογα με τις επιχειρήσεις. Όμως ε, υπάρχουν και αλλαγές ε, όσον αφορά το προφίλ των κρατουμένων ε, υπάρχουν 2.000 άνθρωποι από την Ερυθρέα, υπάρχουν και άνθρωποι από τη Σομάλια. 70% περίπου λοιπόν είναι άνθρωποι ε, που προκαλούν ε, ανησυχίες σε, στην ύπατη αρμοστία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκενωθούν έτσι ε, απλά. Επιστρέφουμε του ανθρώπους που επιθυμούν να επιστρέψουν. Μιλάμε για 15.000 ε, ανθρώπους φέτος που έχουν ωφεληθεί από αυτό το ε, σύστημα που ε, ξεκίνησε με πρωτοβουλία και υπό την αιγίδα της Task Force που συνέστησαν ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση. Εθνικότητες. Νίγηρα, Σιρέρα Λιώνα, ε, Γκάνα, Υποσαχάρη Αφρική, αλλά και Πακιστάν, Μαγκλαντές. Επίσης, υπάρχουν και μετανάστες που δεν βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, αλλά επιθυμούν να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Ξέρετε ότι η ε, Λιβύη ε, είναι χώρα υποδοχής άνω των 600.000 μεταναστών. Η κατάσταση λοιπόν είναι αρκετά περίπλοκη. Ε, γι' αυτό και ε, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με όλες τις κατηγορίες μεταναστών που θέλουν να επιστρέψουν. Επίσης, από τη Σάμπα ε, ξεκινήσαμε επιχειρήσεις εκένωσης από τον νότο της χώρας και επιστρέψαμε πολλούς μετανάστες στο Λάγος. Το θέμα τώρα είναι πώς θα χειριστούμε από εδώ και πέρα την κατάσταση ε, με τους ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται στα, κράτη, στα κέντρα κράτησης. Προσπαθούμε με ε, τη Λιβύη να ανοίξουμε ε, ασφαλείς στέγες μεταναστών, ιδίως για τους, για τους εξαιρετικά ευάλωτους μετανάστες. Έχουμε το παράδειγμα μιας εγγύου μητέρας η οποία θα επιστραφεί, σύντομα. πέρασε κάποιες εβδομάδες σε ένα τέτοιο ε, σε μια τέτοια ασφαλή στέγη και θα επιστρέψει σύντομα στο Μαλί. Επίσης, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και την δυναμική ε, στην αγορά εργασίας που επικρατεί στην ε, χώρα. Ξέρετε, 600.000 άνθρωποι βρίσκονται στη χώρα, μετανάστες, και εργάζονται οι περισσότεροι, ακόμη και αν εργάζονται παράνομα. Γι' αυτό και είναι και αυτή μια διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι και η επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορούν να συμβάλλουν και αυτή στην ε, σταθερότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω τώρα από τον εκπρόσωπο της ε, ε, επιχείρησης διάσωσης και μάλλον βοήθειας και διάσωσης στην Μεσόγειο από είστε από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Αυτή τη στιγμή θέλουμε τα βασικά σημεία και είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι πολλά ε, θα, θέματα θα προκύψουν και αργότερα στη διάρκεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες διαφάνειες που πιστεύω θα βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να παρακολουθούν ε, την κίνηση στην κεντρική, ανατολική και δυτική Μεσόγειο. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το παρατηρείο για την έρευνα και τη διάσωση στη Μεσόγειο. Η μετανάστευση αυξάνεται ε, προς αυτές τις όλες τις πλευρές γιατί έχουν κλείσει τα λιμάνια της Ιταλίας και της Μάλτας. Μετά από τη Μάρεν Όστρομ της Ιταλίας ε, και τη διακοπή της αυτή η δράση ε, έχει γίνει ε, πιο σημαντική ακόμα και ε, υπήρξαν διάφορες καταγγελίες ε, και μάλιστα πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες ε, όσον αφορά την παραβίαση και την συνεργασία των ΜΚΟ με τις, τους διακινητές. Αυτό είναι το υπόβαθρο λοιπόν. Η Σαρομέντ είναι ταυτόχρονα κονσόρτσιουμ αλλά και, μια πλατφόρμα. Είναι ένα κονσόρτσιουμ πολύ ε, διεπιστημονικών ερευνητών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων που εργάζονται στη, σχετικά με τη θαλάσσια μετανάστευση. Τα μέλη μας περιλαμβάνουν τις ΜΚΟ έρευνας και διάσωσας που δραστηριοποιούνται από το 2015 και μιλώ για το παρελθόν γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι ΜΚΟ διάφορες νομικές προκλήσεις και έχουν προβλήματα να μείνουν ε, λειτουργικές. Ε, έχουμε σε Με την, του ε, ε, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, το Σαλβαμέντο Μαρίτιμο Μαριτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα σωρό οργανισμοί Έχουμε και οργανισμούς υπεράσπισης και παρακολούθησης, ε, έχουμε οργανισμούς ε, επίλυσης των διαφορών και έχουμε και ερευνητικά πανεπιστήμια. Η αποστολή είναι να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο έρευνας και διάσωσης ανεξάρτητο με βασικό και μέρημνα την έρευνα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τη συλλογή, αποθήκευση και ανταλλαγή και διάδοση αξιόπιστων στοιχείων, πράγμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα καλύτερα μέσα επίσης ε, ε, τα έχουμε από το Διεθνή Οργανισμό ε, ναυτιλίας, αλλά ε, δεν έχουμε ε, κάποια δικιά μας με βάση δεδομένων. Θέλουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Επιτόπου συνεργαζόμαστε με, με πανεπιστημιακούς και με άλλους φορείς. Η μεθοδολογία μας περιλαμβάνει εταίρους ε, στην θάλασσα που συλλέγουν στοιχεία έρευνας και διάστησης μέσω μιας τυποποιημένης έκθεσης, ώστε να έχουμε ομοιομορφία και συγκρισιμότητα στα στοιχεία. Έπειτα έχουμε ε, στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες. Ε, τα, τα, τα, στα στοιχεία μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη. Ε, Όταν τα συλλέξουμε, τα αναλύουμε οι ερευνητές και τα διάφορα διάφορα πανεπιστήμια και διαδίδουμε τα αποτελέσματα μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπως για παράδειγμα ε, την ε, διάφορη βιβλιογραφία. Έχουμε την έκθεση Mare Clausum, ήταν η τελευταία που λέτε έκθεση ε, όπου έχουμε μια πρωτοβουλία στρατηγικής ε, αμφισβήτησης από την Ντίκλαντ όπου καταγγέλλει την Ιταλία και καταφεύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου γιατί λέει ότι συνεργάζεται με τη Λιβύη και η, πρακτική που ακολουθεί είναι η κατεξουσιοδότηση απόθεση στην ανοιχτή θάλασσα. Εδώ έχετε μια εικόνα για την εσωτερική έκθεση για τα κάθε περιστατικό. Αυτό το χρησιμοποιούμε για συλλέγουμε στοιχεία και εδώ έχετε την πρώτη σελίδα του SAROMED όπου θα δείτε και διάφορες άλλες λεπτομέρειες για μας, ποιοι είναι οι εταίροι μας, ε, ιστορίες ε, διάσωσης, ε, έρευνας και διάσωσης από το 15 μέχρι και το 17 και μετά έχουμε και διάφορες, μια ευρύτερη εικόνα για τους κανονισμούς που ισχύουν πάνω στους οποίους βασίζονται οι δραστηριότητές μας. Αυτά είχα να σας πω και αν μου επιτρέπετε οι δύο λεπτά ακόμη, έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να θέσω στους συναδέλφους ε, εδώ στο πάνελ, αν μου επιτρέπετε, για την Ευρωπαϊκή υπηρεσία, νομική υπηρεσία για τις ε, πλατφόρμες αποβίβασης. Είπατε ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν ισχύουν έξω εδαφικά, ακόμα και αν η έρευνα και η διάσωση και η απόθεση στη συνέχεια γίνεται από ευρωπαϊκούς ε, φορείς οι οποίοι λειτουργούν έξω εδαφικά. Διερωτώμε λοιπόν τι κάνετε με την παράγραφο 21 που λέει ότι οι περιστάσεις δεν μπορούν να υπάρχουν να καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρίς να εφαρμόζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή η εφαρμοσιμότητα του ε, ευρωπαϊκού δικαίου υπονοεί και την εφαρμοσιμότητα, την, ε, ότι είναι εφαρμοστέο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Έπειτα, Σύμβαση της Θάλασσας. Ε, θα πρέπει να υπάρχει δέουσα επιμέλεια και το καθήκον σε διάσωση, άρθρο 88, αυτό είναι εγγυημένο μέσω νομικής δράσης και επιχειρησιακών δράσεων. Δεύτερη ερώτηση, τι σημαίνει διάσωση. Γιατί η Λιβική Ακτοφυλακή κάνει διάφορες ε, δράσεις, αλλά στην ουσία σημαίνει ε, ε, αυτό που κάνει είναι απαγόρευση και πιθανές αποβιβάσεις. Το είδαμε το Νοέμβριο τώρα, όπου 19 άνθρωποι προέρχονταν από διάφορες χώρες, Ερυθρέα, Σομαλία και Σουδάνα, που είναι επικεφαλής ε, στην ζήτηση ασύλου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ε, αναγκαστικά ε, αποβιβάστηκαν στη Μισράτα, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα στην αποβίβασή τους. Η Λιβύη θεωρείται ασφαλής χώρος, ασφαλής χώρα όσον αφορά τις νομικές προδιαγραφές που ισχύουν και το καθεστώς έρευνας και διάσωσης ή ακόμα και για άσυλο θα χρειαζόταν ένα επιχειρησιακό MRCC κατά τη γνώμη μου που να μπορεί να αντιδράσει στις ε, περιπτώσεις ε, MICC και SAR. Ε, η Λιβύη δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες περιστάσεις. Η Λιβυκή ακτοφυλακή είναι γνωστή για βία άσκηση βία στη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνα και διάσωση. Το ανέφερα ήδη στι 20 Νοεμβρίου, ήταν το τελευταίο γνωστό περιστατικό. Εφόσον δεν υπάρχει πλαίσιο και μηχανισμός ε, για την εξυπηρέτηση αυτής ε, της ε, περιφέρειας, πώς, πώς θα γίνει λοιπόν αυτό για την EIS, η πρόσθεση σας για την αλλαγή της πολιτικής αποβιβάσεων. Εσείς έχετε συστήσει μια πρόταση την οποία παρουσιάζεται 15 Νοεμβρίου που έχει στόχο να σταματήσει τις αποβιβάσεις στην Ιταλία μέσω του τέταρτου κανόνα που περιλαμβάνεται στο, εφαρμοσ... στο ισχύον πλαίσιο, το RCC θα αποφασίζει κάθε φορά. Ισχύει όντω αυτό ότι δηλαδή είτε η Λιβύη είτε την Ισία, που είναι μάλλον οι δύο χώρες που θα μπορούσαν ενδεχομένω να είναι σε τέτοια θέση, να θεωρηθούν ασφαλείς για την ε, αποβίβαση μέσα στο κατά την άποψη e της ε, e IOS και στο IOM αναφέρατε ότι ο μηχανισμός εθελοντικής κράτησης, τον οποίο αναφέρεστε, ναι, ναι, τελευταία μου ερώτηση μάλιστα. Στην ουσία εστιάζει στο να επιστρέφουν οι άνθρωποι στην χώρα τους. Αν όμως τηρούν τα κριτήρια για το άσυλο. Πού επιστρέφονται. Είπατε για τον Νίγηρα, είπατε για άλλες χώρες ότι τα προγράμματα έχουν τελειώσει. Ακριβώς τι κάνετε με ανθρώπους που πρέπει να προστατευθούν. Α, αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θα μπορούσατε να απαντήσετε τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Σπινέλη. Μπάρμπαρα. Μετά Κορνίλια Ένστ. Stevens, Sargentini. Μπάρμπαρα Σπινέλη ξεκινάει. Difficile intervenire visto che le είναι δύσκολο να παρέμβουμε γιατί τα πιο σημαντικά ερωτήματα που ήθελα και εγώ να θέσω τα ε, υπέβαλε η Βιολέτα Μορένο Λάξ, την οποία ευχαριστώ και ε, για το έργο της με την ΣΑΡΟΠΜΕΤ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους θεσμούς που εκπροσωπούνται εδώ να εγκαταλείψουν ε, τα την υποκρισία, το διπλό λόγο που χρησιμοποιούν ε, όταν μιλάνε για αυτούς τους ανθρώπους και να δούνε με ρεαλιστικό τρόπο τις τραγωδίες που εκτελήσονται στη Μεσόγειο. Να γνωρίσουμε ε, κυρίως ότι είμαστε ενώπιον μιας τεράστιας αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών θεσμών. Η Κομισιόν ε, πέρεται για τη μείωση των ε, αφήξεων, αλλά όχι ε, για τον παράλληλα αυξημένο αριθμό θανάτων στη θάλασσα. Δεύτερον, η ζώνη έρευνα και στη Λιβύη, το ανέφερε όντως η Βιολέτα, και η βάση δεδομένων του Διεθνού Οργανισμού Ναυτιλίας είναι μια ζώνη ΙΣΑΡ που δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Γενέβης, γιατί δεν έχουν πολιτική ασύλου, γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες να κάνουν έρευνα και διάσωση και άρα δεν κάνουν στην πράξη έρευνα και ε, διάσωση. Άρα λοιπόν διερωτώ με μήπως είναι σκόπιμο να καταργηθεί η ζώνη ΣΑΡ της Λιβύης και η εκένωση. Οι απαντήσεις που λάβαμε από τον υπατερμοστία του ΟΗΕ είναι ότι ακόμα δεν μπορεί να ανοίξει δικό του κέντρο ε, εκένωση ότι κάποιοι μετανάστες έχουν φτάσει προς τον Ήγηρα και ότι εν πάση περιπτώσει οι πανεπατρισμοί αυτού του τύπου λειτουργούν μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση σεβαστεί τις δεσμεύσεις επανεγκατάστασης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σέβεται τις αποφάσεις περί μετεγκατάστασης. Οι φυλακές στην νομική άποψη παρουσιάζονται πλέον σαν κάτι το φυσιολογικό. Αυτά έχω να πω γιατί πιστεύω πως οι συνάδελφοι έχουν και άλλα να πούνε σχετικά. Α, ναι, και κάτι τελευταίο. Έκανα μια ερώτηση στο όνομα της ε, κυρίας Βεριζιά προς την Κομισιόν. Έγινε ε, λοιπόν μια προφορική ερώτηση και θέλω να ακούσω μια απάντηση της Επιτροπής σήμερα, όχι κάποτε. Από τον Φιλίππο Γκράντι ακούσαμε την απάντηση, από την Κομισιόν τίποτα. Να επιστρέψω και πάλι στον κύριο Βίνο. Για να το θέσουμε το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ έχει μπει στον να θέσει το θέμα αυτό. Θα επιστρέψουμε στο θέμα λοιπόν. Η κυρία Κορνίλια είναι τώρα έχει το λόγο. Κορνίλια. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την τελευταία ομιλήτρια γιατί μα μίλησε μέσα στην καρδιά μα τρεις παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχάς, κάποια στιγμή, κάποια μέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εδώ οι εκπρόσωποι της που βρίσκονται εδώ, μήπως κάποια στιγμή θα ντραπούν, δεν ντρέπονται, που έρχονται και μας λένε αυτά που μας λένε. Μας τα παρουσιάζονται αυτά σαν αξιοπρεπή πράγματα ντροπή. Λίγο ηθική να υπάρχει, πέρα από τις ανοησίες που μας λέτε. Είμαι πραγματικά ε, αγανακτισμένη. Είναι ντροπή και όνειδος αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλους όσοι σας ακούνε, μας περνάτε για χαζούς. Τέτοιες προσεγγίσεις που τις παρουσιάζονται για ανθρωπιστικές. Αυτό το σύστημα της μη επιστροφής, πώς θέλετε να το εφαρμόσετε με τις πλατφόρμες αυτές, με τα συστήματα αυτά. Κατά δεύτερον, θέλω να ξέρω και θα ξέρετε σίγουρα πώς δρούν οι ακτοφύλακες ε, όταν ε, υπάρχει ένα καράβι στη θάλασσα από γειτονική χώρα. Το ξέρετε ότι λαμβάνω χώρα βασανιστήρια. Ότι πνίγεται ο κόσμο στη θάλασσα γιατί κάθονται και του κοιτάνε. Τρίτο που ήθελα να πω. Είπατε ότι τα ελεγχόμενα κέντρα δεν υπάρχει θέμα γενική ε, ε, σύλληψη κτλ. Πώ θέλετε να εξηγήσετε όλα αυτά, με ποια βάση λοιπόν βασίζεστε. Αυτά ήθελα να μου πείτε πέρα από το γεγονός ότι και εγώ Ντρέπομαι για αυτό που αντιπροσωπεύετε εδώ. Um, Συνάδελφοι, να επενθυμίσω απλώς ότι σε 10 λεπτά ε, θα φύγουν οι διερμηνείς μας. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο για να λάβουμε τις απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις που θέσατε εσείς και η κυρία Μορένο Λάξ. Κυρία Στίβενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συναδελφοί, να σας ε, παραπέμψω σε μία έκθεση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και στείλαμε μία απάντηση στην τελευταία άμα, χώρα για μετακόμιση στη Μεσόγειο. Και είδα, λοιπόν, τη σχετική αναφορά στη νομική στην έκθεση τη νομική υπηρεσία. Θα πρέπει λοιπόν οι μετανάστε και οι πρόσφυγε να μεταφέρονται σε ένα ασφαλέ μέρος, σε μια ασφαλή τοποθεσία. Αυτό δεν έχει οριστεί όμω ε, επαρκώ. Μεταξύ, των, μεταξύ άλλων, να μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να του πηγαίνουν του μετανάστες σε τρίτε χώρε. Είναι εντελώ παράνομα. Αν είχαμε τέτοιες συμφωνίες με όλες τις χώρες ε, με όλες τις χώρες της Μεσογείου δεν θα υπήρχαν πνιγμοί πλέον. Και αν γινόντουσαν αυτά, δεν θα υπήρχαν άμα, ε, ε, θάνατοι. Αλλά η Ευρώπη προτιμάει να ασκεί την πολιτική των ελεύθερων συνόρων. Όποιο θέλει μπορεί να μπει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να οργανώνουμε μια σωστή ε, υποδοχή των ανθρώπων αυτών σε τρίτες χώρες, προκειμένου να μην χάνουν ζωές και να υπάρχει ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ. Είναι κρίμα που δεν είναι δημόσια η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, γιατί όταν τη διαβάζει κανείς ε, μπορεί να κατανοήσει και διάφορες διαστάσεις του θέματος. Αυτό που μου λείπει είναι η βασική παραδοχή ότι αν υπήρχαν ασφαλείς λιμένες και καταφύγια στην Βόρεια Αφρική, φυσικά και δεν θα διαφωνούσε κανείς με την αποβίβαση ανθρώπων, αλλά εννοώ πραγματικά ασφαλή καταφύγια, με ένα σύστημα ασύλου το οποίο θα λειτουργεί και θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Δεν νομίζω πολλοί να διαφωνούσαν με κάτι τέτοιο. Όμως, μπορείτε... Ε, όσο και να την να ψάξετε την ε, πρόταση της Κομισιόν, όσο και να θέλει κανείς να την εξοραίσει, δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τέτοια ασφαλή καταφύγια ε, στη Βόρεια Αφρική. Και θεωρώ πολύ προβληματικό στην περίπτωση αυτού του πλοίου υπό σημαία Παναμά, Παναμά που βρέθηκε στη Μισράτα και από την οποία έγινε βίαιη αποβίβαση των ε, επιβενών μεταναστών. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό και επικίνδυνο. Διότι τα εμπορικά πλοία που δεν βρίσκονται υπό ευρωπαϊκή σημαία θα μπορούσαν να παρακάμπτουν τους κανόνες. Γιατί τους είπαν ε, οι οι κάτοχοι αυτού του πλοίου λόγω του γεγονότος ότι βρίσκονταν υπό σημαία Παναμά, ότι πηγαίνουν στη Μάλτα και τελικά κατέληξαν να ξεφορτώνουν αυτοκίνητα και αυτούς στην Μισράτα. Εδώ είναι, πρόκειται για ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, με συγχωρείτε κύριε, αλλά νομίζω ότι δεν έχετε ακριβώς καταλάβει την ε, διαφορά ανάμεσα στο τράφικινγκ και το λαθρεμπόριο. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι που επιδίδονται και στις δύο δραστηριότητες, αλλά θα πρέπει να γίνεται διάκριση. Όταν μιλάτε για τράφικινγκ και στην πραγματικότητα αναφέρεστε στο λαθρεμπόριο, τότε νομίζω ότι η, συζήτηση μαζί σας θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Οι ορισμοί είναι πραγματικά πολύ σημαντικοί ε, σε αυτή την ε, συζήτηση. Για το Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης. Ε, είχαμε μια κλεισμένα των θεωρών συνάντηση με την ύπατη αρμοσία τον Σεπτέμβριο, όπου ήδη είχα εκδηλώσει τις ανησυχίες μου για το γεγονός ότι τίνεται χείρα βοηθείας στο Συμβούλιο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των κέντρων αποβίβασης. Και επισημαίνω για άλλη μια φορά ότι υπάρχει και επιστολή του Υπουργείου μου από την Ολλανδία για τη συνεργασία που έχουν με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστασης για την ολοκλήρωση αυτών των κέντρων. Ενώ εμένα μου είχατε δώσει την εντύπωση το Σεπτέμβριο ότι και εσείς είχατε εκπλαγεί από αυτό τον εφιάλτη που πρότεινε το Συμβούλιο για τη δημιουργία αυτών των ε, κέντρων αποβίβαση. Νομίζω ότι δεν συνάδει με την αποστολή ε, του ΟΗΕ ούτε του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αυτή η δραστηριότητα. Και τελικό ερώτημα. Υπάρχει τρόπιμα, τρόπος να καταστεί δημόσια η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι απόρριτη. Πρόεδρος, ε, προειδοποιώ απλώς ότι θα συνεχίσουμε στα αγγλικά για τις απαντήσεις γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Dietmar Köster. Ευχαριστώ, Κλόντ. Νομίζω ότι αποτελεί ένδειξη περιφρόνησης της Επιτροπής όταν παρουσιάζονται ε, τέτοιες εκθέσεις εξοραϊσμού της κατάστασης εδώ στην Επιτροπή μας. Στις 20 Νοεμβρίου στον Ιβίν το πλοίο το εμπρευματικό βρίσκονταν μετανάστες μπροστά στις ακτές της Λιβύης και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο παρά τη θέλησή τους. Ερώτησή μου προς τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση. Εσείς δεν είχατε τη δυνατότητα να βρίσκεστε εκεί για να, εξασφαλ... την ασφάλεια των μεταναστών. Έχετε διατηρήσει επαφές με τους ανθρώπους αυτούς. Ξέρετε να μας πείτε τι συμβαίνει και που βρίσκονται. Δεύτερον, γνωρίζετε ότι τακτικά ε, πεθαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα κέντρα κράτησης στη Λιβύα. Έχετε στοιχεία για τις αιτίες θανάτου, για τον αριθμό των θανόντων. Ποιο συλλέγει τους, ε, τους αριθμούς, αυτά, τα αριθμητικά αυτά στοιχεία και με ποιες πηγές. Πρόεδρος, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Λυπάμαι που έχουμε χρονικό ε, περιορισμό. Αλλά δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Η κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ, Κλόντ. Τρει ερωτήσει έχω να κάνω. Και εγώ από πλευρά μου, εν συντομία και πολύ συγκεκριμένα, στα ενίδια του τρει σε ό,τι αφορά τον αριθμό των 34.000 ε, ατόμων που εκενώθηκαν. Είπατε ότι αυτό είναι πρόοδος. Εξ όσων γνωρίζουμε εμείς, πέρα από αυτόν τον αριθμό, έχουμε και 600.000 επιπλέον άτομα σε κέντρα και εκτός κέντρων. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ αποκλίνοντα, 60.000 ή 34.000, άρα δεν έχει γίνει πολλή δουλειά. Η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης τώρα. Δεν εχει γινει πολλη δουλεια η ποινικοποιηση τη αλληλεγγυη τωρα δεν μπορουμε να το κάνουμε αυτό. Στην αλληλεγγύη. Όλοι αυτοί οι λόγοι που απαριθμούνται και άλλες παραβιάσεις Δυστυχώς αυτό επηρεάζει τη θεώρηση του φαινομένου και την αντίληψη περί αλληλεγγύης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ΜΚΟ και αυτά που μας καταγγέλουν για τους διακινητές, έχετε αποτελέσματα για το γιατί κάνουμε γενικές διατυπώσεις για το θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται τόσο γενική διατύπωση. Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε, Σεσίλ. Και τέλος ο κύριος Γιούρεκ και μετά θα ακούσουμε τους πανελίστες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η, προετοιμασία, η προστασία συγγνώμη, των συνόρων περιορίζεται και από το εθνικό δίκαιο και είναι τμήμα του κράτους δικαίου. Δεν είναι δυνατόν να μην σέβεται τον νόμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πίεση για να καταργηθούν τα σύνορα σε καιρού ανθρωπιστική κρίση που μιλάμε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια σημαίνει να σεβόμαστε τον νόμο. Να σεβόμαστε τον νόμο των άλλων, τον νόμο της οικογένειας, της κοινωνίας. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό, αυτή η κρίση θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από δηλώσει Ευρωπαίων πολιτικών που ενθαρρύνουν να λαμβάνονται τέτοιε επικίνδυνε αποφάσει για τη μετανάστευση. Το πρόβλημα λοιπόν θα ήταν πιο μικρό στο μέλλον. Αν... Και αυτό, αν ήταν το, πρόγραμμα, το πρόβλημα αυτό πιο περιορισμένο, θα μπορούσαμε να δώσουμε πραγματική βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να φεύγει από τα σπίτια του, να κάνει τακτική μετανάστευση. Δεν κρίνω αυτός που πήραν το λόγο, απλά προσπαθώ να ενθαρρύνω την εξέβρεση λύσεων και να περιορίσω και τα προβλήματα που υφίστανται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα ζητήσουμε από τους συναδέλφους να απαντήσουν ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Κανείς δεν ε, θέλει να σας δυσαρεστήσει. Να είσαστε πραγματικά άδεκτοι, γιατί μιλάμε για τη Λιβύη. Έχω μεταβεί και εγώ στη Λιβύη και οι πολλοί από τους συναδέλφους έχουν δαπανίσει χρόνο και ενέργεια, ξέρουν γιατί μιλάνε, έχουν μελετήσει καλά τα ζητήματα αυτά. Έτσι λοιπόν να τα λάβατε αυτά και προσπαθήστε να απαντήσετε τα βασικά σημεία. Και στο σημείο αυτό η διερμηνία